Αγαπητοί συνάδελφοι, σα ζητώ να καθίστε στι θέσει σα, ούτω ώστε να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μα και θα περάσουμε στο σημείο 14 της ημερήσια διάταξη, και θα ήθελα να καλωσορίσω την Έλκε Κένιγκ, πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην Επιτροπή μας το 2017 στην Επιτροπή μας και είναι εδώ για να παρουσιάσει την ετήσια έκθεση 2016 του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Και θα έχουμε και την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις επίσης για πρόσφατες περιπτώσεις εξυγίανσης στην Ευρώπη και που έδειξαν την ικανότητα του μηχανισμού, του πλαισίου αυτού εξυγίανσης που δεν είχε δοκιμαστεί να δράσει ε, αποτελεσματικά σε διάφορες περιπτώσεις μέσα στα πλαίσια των κανόνων μας και να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Είναι ένα θέμα συζήτησης και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κόνιγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί βουλευτές, με μεγάλη μου χαρά σήμερα θα σας μιλήσω για να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεσή μας για το 2017. Επίσης δημοσιεύεται αυτές τις μέρες Οπότε και μπορώ να σας ε, δώσω κύριε Πρόεδρε ένα αντίγραφο αυτής. Αλλά φαντάζομαι ότι ενδιαφέρεστε περισσότερο για το μέλλον και για τα τρέχοντα ζητήματα παρά για το παρελθόν. Αυτό θα προσπαθήσω να σας ε, αναπτύξω. Οπότε θα πρέπει να βελτιώσουμε την ετοιμότητα και την εξυγίνηση των περίπου 140 τραπεζών για τα οποία έχουμε την εντολή ήταν και είναι ακόμα βασική μας προτεραιότητα και βασικός σκοπός του ε, ενιαίου Σύμβουλου αλλά για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό σε έναν χρόνο δεν είναι εφικτό, αλλά, αλλά μας βοηθούν οι εθνικές αρχές εξυγίανσης με, με τον μηχανισμό εξυγίανσης, ε, με αυτά τα προγράμματα ε, του 2016 και αυτά τα 92 προγράμματα τα οποία καλύπτουν τις περισσότερες, περισσότερους ομίλους τους τραπεζικούς της Τραπεζικής Ένωσης. Και είπαμε ότι αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε ενημερωμένα δεδομένα της τράπεζας και όσον αφορά την δομή του παθητικού των υποχρεώσεων της τράπεζας το 2016 ζητήσαμε από τις τράπεζες να μας δώσουν αυτά τα δεδομένα του παθητικού των υποχρεώσεών τους με ε, κάποιες συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό το κάναμε σε συνεννόηση με τον ΙΕ, υποπτικό μηχανισμό, ούτω ώστε να μην έχουμε επικάλυψη για τι ε, αιτήσει δεδομένων που βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών. Αλλά είπαμε ότι οι υποπτικέ αρχές δεν συλλέγουν σε τακτικά διαστήματα αυτά τα δεδομένα. Οπότε ο στόχος αυτών των δεδομένων είναι το ότι θέλουμε να δούμε εάν καλύπτονται οι βασικές προϋποθέσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις, το MREL, αλλά επίσης είπαμε ότι είναι απαραίτητα κατεπηγώντας αυτά τα δεδομένα ούτω ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι αποφάσεις μπορεί να πάρουμε όσον αφορά την ε, εξυγίανση για διάθεση κάποιες τράπεζες. Το 2016 έχαμε εγκρίνει ε, σαν μια προπαρασκευαστική, προκαταρική προσέγγιση στο MRAL, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Και αυτό το νομοθέτημα συνεχίζει να εξελίσσεται. Πρόκειται για αυτή τη δέσμη μέτρων του Νευρίου που θα, τότε πρόκειται να ολοκληρωθεί. Αυτή η δέσμη μέτρων ε, καλύπτει τα προαπαιτούμενα του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος σε σχέση με την οδηγία για εξηγήνωση των ε, τραπεζών όσον αφορά τις ε, ζημίες. Ε, και είπαμε ότι το MRL θα πρέπει να ολοκληρωθεί, μια που χρειάζεται ξεκάθαρο τοπίο για τις τράπεζες. Και θα πρέπει τώρα να δούμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί αυτό το σύνολο κανόνων. Αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο Επομένως θα έχουμε τώρα μια ιεραρχία για τους πιστωτές και επίσης για την επιλεξιμότητα. Αυτό πάντοτε αφορά τις τράπεζες και είπαμε ότι δεν υπάρχει λόγος κανείς να τηρεί στάση αναμονής. Οι τράπεζες προσπαθούν να αποφύγουν κάποιο είδους ε, διάσωση που θα έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορολογουμένους. Ε, και πέραν του τι είναι το 2016, προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε κάποιους στόχους μη δεσμευτικούς για τα ε, MRL και επίσης ε, τις προσδοκίες μας τις γνωστοποίησαμε στις τράπεζες οπότε και οι τράπεζες άρχισαν να προσανατολίζονται προς εκείνους τους ε, στόχους. Στο βαθμία Βεβαίως και αυτού του είδους ο προγραμματισμός εξυγένσης δεν περιορίζεται στα MRL. Ε, έχουμε και άλλες ε, σημαντικές λειτουργίες, πρόσβαση ε, στις υποδομές των χρηματαγορών και αυτά επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε να δούμε τι παραθυράκια υπάρχουν στο νομικό πλαίσιο από πλευράς άλλων οργανισμών, γιατί πρόσφατα δεν είναι μια απλή δομή, είναι ένας λαβύρινθος οι ρυθμίσεις και όπως σας είπα ο προγραμματισμός της εξυγίωσης δεν μπορεί να κληρωθεί μέσα σε μια χρονιά. Η δε συνεργασία με τις εθνικές αρχές διάσωσης είναι πάρα πολύ σημαντική ούτως ώστε να υπάρχουν πολιτικές οριζόντιες και οι άρεστες πρακτικές να ε, διαδίδονται. Και το 2016 είπαμε ότι έχουμε προχωρήσει όσον αφορά το ενίο Ταμείο Εξυγίανσης και φέτος είχαμε 6,6 εκατομμύρια συγγνώμη δισεκατομμύρια ως συμβολή και τώρα το Ταμείο έχει στη διάθεσή του σχεδόν 17,4 δισεκατομμύρια οπότε και όπως ε, είπαμε έχουμε συνάψει συμφωνίες διαμικής διευκόνησης με τα κράτη-μέλη οπότε και βοηθούμε το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει για να υπάρχει ε, κάποιο είδους κοινή αντιμετώπιση για το Ταμείο. Τώρα, όσον αφορά το 2017 και για την περίοδο μετά το 2017, για όλους αυτούς τους τομείς που είπαμε, προσπαθούμε να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε την δραστηριότητά μας, προσπαθούμε να έχουμε λειτουργικά ε, προγράμματα διάσωσης, να εξασφαλίσουμε ότι στον πραγματικό κόσμο αυτά αποδίδουν, λειτουργούν και θέλουμε να υπάρχει ιεραρχία του τι γίνεται στην ε, εξυγίανση, να δούμε ε, οι ζημίες πώς ε, αποδεικνύονται και να δούμε τι ισχύει όσον αφορά τις εταιρείες και το εταιρικό δίκαιο. Οπότε πώς τι με τις στρατηγικές της εξυγίανσης έχουμε αρχίσει να ασχολούμεθα με κάποιου πρακτικές τροχοπέδες και αυτό προσπαθούμε να έχει τέτοιου είδου χαρακτήρα βαθμιαία. Επίσης να δούμε τι γίνεται με κάποιο είδους ε, διασυνοριακά, διαμετριακά φαινόμενα ε, και γι' αυτό και κάνουμε κάποιες ασκήσεις επί χάρτου, κάποιο είδους προετοιμασία στην Τραπεζική Ένωση και έχουμε άλλες προσκευές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη της Τραπεζικής Ένωσης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε κάποιες ε, τριμερείς τέτοιες συναντήσεις με ΙΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Ο στόχος μας τώρα όσον αφορά τους στόχους MRL, το είπαμε επανειλημμένα, ότι είναι το ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε κάποιους δεσμευτικούς στόχους για όλους τους τραπεζικούς ομίλους και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δούμε από πλευρά ποιοτική τι γίνεται με τα MRL εσωτερικό των ομίλων. Να δούμε ποιο είναι επιλέξιμο σε αυτά τα πλαίσια και έτσι να βασίζουμε κάθε απόφαση ε, στην ισχύουσα νομοθεσία παρακολουθώντας την δέσμη μέτρων του Νοεμβρίου όπως εξελίσσεται. Δεν είναι εύκολο το έργο μας, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία και βεβαίως θα λάβουμε υπόψη τις πρόσφατες εμπειρίες με τις ε, περιπτώσεις ε, εξυγίανσης όπως ξέρετε τι, τι έγινε τις τελευταίες εβδομάδες. Στις 7 Ιουνίου το Ταμείο Διάσωσης ενέκρινε ε, την πρώτη εξηγήνση με απόφαση που πυροδότησε την πώληση της Banco Popular στην Banco Santander για ένα ευρώ. Η δε ε, υπηρεσία διάσωσης και εξηγήνσης της Ισπανίας έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος διάσωσης και εξηγήνσης Μπορεί να πει κανεί ότι αυτό ήταν σαν υπόθεση κλασική σχολικού εγχειριδίου ε, στα πλαίσια της οδηγίας BRRD ε, αλλά υπήρξε στενή συνεργασία εθνικών αρχών με τις ευρωπαϊκές ε, αρχές. Τρίτη βράδυ με Τετάρτη πρωί κλείσαν αυτές οι συμφωνίες και έγιναν τα σχετικά Μια εβδομάδα πριν είχε ξεκινήσει η διαδικασία στο εργό της τράπεζας και στη συνέχεια είχαμε τη διαδικασία πώλησης στον ιδιωτικό τομέα και το ενιαίο συμβούλιο μπόρεσε πάνω σε αυτό να στηριχτεί. Δεν θα μπορούσαν αυτά να γίνουν βέβαια από το βράδυ ως το πρωί αν δεν είχε προετοιμαστεί αυτή η διαδικασία. Τώρα η κατάσταση των δύο μικρών ε, Ιταλικών τραπεζών στην περιοχή του Βένετο την τράπεζα Βιτσέντζα και την Φινιμπάνκα ε, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν προβληματικές και αφαιρέγγιες ε, στις 23 έκτου. Διάφερε αυτή η περίπτωση, διότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπήρχε διασύνδεση, υπήρχε συρρήκνωση από πλευράς ε, αυτής της διασύνδεσης και του μεγέθους και η μόνη τους λειτουργία, η πιο σημαντική δηλαδή οι καταθέσεις και αποταμιεύσεις ε, διετίθετο από 30 άλλες τράπεζες στην περιφέρεια αυτή. Οπότε το Συμβούλιο Διάσωσης κατέληξε το ότι η διάσωση δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον για την κάθε τράπεζα και για μαζί, οπότε θα μπορούσαν, όπως προβλέπεται στο κοινωνικό κανονισμό, να ενταχθούν στην συνήθεια ε, πτωχευτική διαδικασία του Ιταλικού δικαίου, χωρίς να υπάρχει για τις ε, αγορές κάποιος κίνδυνος ή για την Ιταλική οικονομία. Οπότε και οι Ιταλικές αρχές απεφάσισαν να ενεργήσουν και την περασμένη εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την άδεια για κάποιο είδους προληπτική κεφαλαιοποίηση της Μοντεπάσχη Σιένα. Και αυτά έγιναν για πρώτη φορά ε, αυτά όλα προβλέπονται βέβαια από την ε, οδηγία για την εξηγένση. και όλα αυτά επαναλαμβάνω ρητός προβλέπονται στην οδηγία για την εξήγηση των τραπεζών αυτά τώρα το, η πρώτη απόφαση που ήταν για την Banco Popular απέδειξε το πόσο το πλαίσιό μας είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό όμως επισημάνθηκαν κάποιοι τομείς που περιέχονται βελτίωση Οπότε ακόμη εξελίσσεται την κατάσταση και ξέρω τώρα είναι νεκροψία της τράπεζας και υπάρχει αυτού του είδους το εργαλείο αναστολής εκροής στην Ισπανία και είπαμε ότι αυτού του είδους το moratorium tool παρουσιάζει πάρα πολλά πλέον εκτίματα όσον αφορά την χρήση του από την αρχή διάσωσης. Τώρα είπαμε όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, ε, βέβαια και αυτή η εξηγένση απέδειξε ότι υπήρχε στενή συνεργασία και το πόσο σημαντικό είναι να αυτά τα δεδομένα για τις υποχρεώσεις τράπεζας θα πρέπει να διατίθενται αμέσως. Και είπαμε επίσης ότι θα πρέπει οι τράπεζες να επενδύσουν όσον αφορά τις δομές τους και την δυνατότητά ε, τους και αυτό ήταν το μάθημα το οποίο αντιλήθηκε. Και τώρα ένα άλλο ζήτημα το οποίο ανέκυψε και δεν είναι βέβαια ούτε αυτό καινούριο. Είναι το ότι σε περίπτωση εξυγίανσης είναι το θέμα της ε, ταμιακής ζωής ή της χρηματοδότησης. Στην Banco ποπολαρ δεν πήγαν καλά τα πράγματα, ούτε αυτή η ρευστότητα υπήρχε. Οπότε, για να αποκατασταθεί αυτή η ρευστότητα την Τετάρτη το πρωί ε, αυτό ήταν πολύ σημαντική ενέργεια και ευτυχώ αυτοί που εξαγόρασαν την τράπεζα μπορούσαν να το κάνουν κατά τα άλλα όμως παραμένει πρόβλημα η χρηματοδότηση τη εξυγίανση, ιδίω όσον αφορά τι πιο κεντρικέ τράπεζε. τώρα η συνεργασία στο ιστορικό τη Τραπεζικής Ένωση είναι και αυτό σοβαρό ζήτημα Εν προκειμένου πάντως επρόκειτο για κάποια θηγατρική αμερικανική. Οπότε η διαμεθοριακή συνεργασία αντιμετωπίστηκε και ήμασταν τυχεροί γιατί όλα αυτά έγιναν με τρόπο θετικό και τελευταίο αλλά σημαντικό. Μπορώ να πούμε γενικώ ότι θα πρέπει όταν κανείς εξετάζει διάφορα συστήματα θα πρέπει κανείς να εξετάζει τι κίνητρα υπάρχουν. Και για μένα η λύση του ιδιωτικού τομέα είναι πάντοτε η καλύτερη, προσφέρει τα περισσότερα πλεονεκτήματα. Αυτή είναι προτιμητέα. Η δάλος, εντάξει, ας γίνει εξυγίανση, αλλά ίσως καταστεί προβληματική όταν έχουμε κάποια αφαιρεγγιότητα η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερο deal για τους πιστωτές. Έχουμε και την σχετική αναγένωση του 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να αξιολογηθεί. Θα πρέπει να δούμε εάν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά αυτό το πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για την εξηγήνωση του... Φτάσαμε τώρα Ιούλιο του 2017. Σα είπα, δεν κάλυψα τα πάντα, αλλά εδώ θα βάλω μια τελεία, γιατί έτσι καλώς έχω μακρηγορήσει και συμπαθάτε μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και για τα θέματα και το πρόβλημα της ρευστότητας των τραπεζών που είναι σημαντικό θέμα που σχετίζεται με το θέμα της στήριξης και νομίζω ότι η Επιτροπή είναι πάρα πολύ προσεκτική για τις περαιτέρω αλλαγές στους ε, κανόνες τους οποίους θα πρέπει να προσαρμοστούν οι φορείς της αγοράς. Αμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και εσάς για τις πρέπει Να μιλήσουμε πάντα για το μέλλον και συμφωνούμε ότι κάποιοι από τους στόχους της ε, Τραπεζικής Ένωσης θα πρέπει να τους προσέξουμε για το μέλλον, γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το χρήμα των φορολογουμένων για να σωθούν οι πτωχεύουσες τράπεζες. Και ε, έχουμε επίσης έτσι ε, κατάτμιση της αγοράς για να δούμε πώς θα θωρακίσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Είπαμε τι έγινε με την εξηγήνση της Banco Popular και των Ιταλικών τραπεζών, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία εφαρμογή το, του πλαισίου που να μην είναι αυθαίρετη και να δούμε κατά πόσον πληρούνται οι στόχοι της Τραπεζικής Ένωσης και έτσι να σώσουμε τις πτωχεύουσες τράπεζες αλλά χωρίς το χρήμα των φορολογουμένων και έτσι να στηριχθεί μια αγορά με διαφορολογικές ε, μεθόδους διάσωσης για τα διαφορετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα το πρωί ο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας δήλωσε ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Εσείς συμφωνείτε Πρέπει να αλλάξουν τους κανόνες. Και προς τα ποια κατεύθυνση. Πάντως νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε εφαρμογή των κανόνων. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι βεβαίως όταν εξετάζετε τις περιπτώσεις εξυγίανσης της Banco Popular και βλέπουμε ποιοι είναι οι κανόνες της Τραπεζικής Ένωσης. Δεν υπήρξε μετάδοση στην αγορά και οι φορολογούμενοι διασώθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη πλευρά δεν θα έλεγα ότι στην Ιταλική περίπτωση αυτό επιτεύχθηκε πλήρως όταν δείτε από την προοπτική της εξυγίανσης. Η εξυγίανση χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για τις μεγαλύτερες τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση συμπεράναμε ότι δεν ήταν μια τράπεζα η οποία ε, είναι ε, τράπεζα δημοσίου συμφέροντος κατά κάποιο τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, έχει κανείς να κάνει με κανονική πτωχευτική ε, διαδικασία και εκεί έχετε εθνική νομοθεσία διότι δεν έχουν εναρμονιστεί οι νομοθεσίες οι εθνικές και οι αρχές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν δημόσιο χρήμα που θα έπρεπε από την Digicom της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκριθεί. Δεν θέλω ε, να κρίνω την απόφαση της DGCOM αλλά θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα μέσα στο σύνολο του ε, πακέτου και όχι βεβαίως κατά τις θερινές διακοπές. Αυτό ήθελα να πω μιλώντας για κίνητρα. Η η ανακοίνωση της Επιτροπής απαιτεί κατανομή βαρών ε, για τους μετόχους, ε, ε, κοινών μετοχών ε, και προνομιούχων μετοχών, δεν απαιτεί διάσωση με ίδια μέσα και είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί από αυτήν ε, την άποψη. Ούτως ώστε να επιτρέψει κάποια εκαθάριση δεν είναι μη ρεαλιστική αν απαιτείται ούτως ώστε να παρασχεθεί ρευστότητα για να έχει μια εκαθάριση ομαλή συντεταγμένη αλλά εκεί χρειάζεται κάποια ευθυγράμμιση. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει και καθάριση τραπεζών κλείσιμο, να κάνουμε συγκρίσεις. Mm. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι διαφορετικές. Περβάνς Μπέρεντσε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κόνιγκ. Και νομίζω ότι είχατε σημαντική στιγμή στην ιστορία ε, την τραπεζική, την ευρωπαϊκή, το ότι υπήρξε αυτή η πρώτη ε, χρήση των εργαλειών που εκπονήσαμε, ακόμη και αν υπήρξε μια αυστριακή περίπτωση για την οποία έγινε λιγότερος λόγος, και φαντάζομαι ότι δεν είχατε σκεφτεί ότι θα έχετε τρεις περιπτώσεις μέσα σε ένα μήνα. Αλλά βρισκόμαστε τώρα στην ώρα όχι της, του απολογισμού αλλά των διδαγμάτων που θα μπορούσαμε να αντλήσουμε από τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην νομοθεσία μπορούν να κινητοποιηθούν σε στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν κινητοποιηθεί για ένα άλλο σκέλος αυτής της συζήτησης μεταξύ risk sharing και risk reduction. Κατανομή κινδύνου και μείωση κινδύνου. Σόσα είπατε στα στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στη συζήτηση που μπορεί να εξελιχθεί αργότερα δεν νομίζετε ότι το πραγματικό επίγον θέμα και το πραγματικό πρώτο δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε είναι η κατεπίγους ανάγκη να έχουμε backstop, να έχουμε στήριξη. Και διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια ένταση μεταξύ των δύο αυτών σκελών, ε, risk sharing και risk reduction, αλλά έχω την εντύπωση ότι μερικοί θα μπορούσαν να θελήσουν να επιβαρύνουν προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, ε, περισσότερο ΜΡΕΛ, ε, ελάχιστη απέτηση, να μην ενισχύσουμε ε, το πρότιμο, την απέτηση ΜΡΕΛ, αλλά πότε δεν φτάνουμε στο backstop. Εμένα μου φαίνεται ότι διαβάζοντας ε, την εμπειρία με τις τρεις περιπτώσεις που είχατε να εξετάσετε. Ευτυχώς ε, δεν είχατε ε, ε, πρόσβαση σε backstop. Δεν υπάρχει μια αντιστροφή των προτεραιοτήτων και η πραγματική προτεραιότητα σήμερα είναι να υπάρξει το backstop Ευχαριστώ θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε και τα δύο. Χρειαζόμαστε να εργαστούμε για το backstop και η εργασία αυτή έχει αρχίσει και προοδεύει θα λέγατε δημόσια ότι ναι. τώρα είναι κατεπίγους ανάγκη να καταλήξετε για το θέμα αυτό, προτού περάστε σε άλλα θέματα. Ε, προσπαθούμε να έχουμε κάποια ισορροπία, να ε, προδεύσουμε και να μην περιμένουμε για το ένα ή το άλλο. Ε, η εργασία για το backstop έχει αρχίσει. Τεχνικά βρίσκεται στην φάση αμοιβεοποίησης που είναι κάτι το πάρα πολύ περίπλοκο Ε, άρχισε με το Ταμείο, Ταμείο Εξυγίανσης, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε με το backstop και ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, με την MREL, ε, διότι βεβαίως το backstop είναι το τελευταίο, το έσχατο μέσο και θα πρέπει τη τράπεζα να έχει αρκετό διάσωση με ίδια μέσα. Νομίζω ότι θα πρέπει βεβαίως αναφέρεται το LFD, αναφέρατε ένα σωρό άλλα πράγματα, τα, θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ε, εμείς και το Συμβούλιο τελικά ε, θα πρέπει να αποφασίσουμε. Ελπίζουμε να μετακινηθούμε ε, στις θέσεις μας και να μετακινηθεί και το Συμβούλιο. Και η Σουίνμπερν. Α, συγγνώμη, δεν σε είδα. Ναι, είμαι έτοιμη. Ναι, νόμιζα ότι θα κάθεσαι απέναντι. Συγγνώμη. Ε, κυρία Κόνιγκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ να αφιερώσετε χρόνο σε εμά σήμερα. Θα ήθελα να επανέλθω στην ισορροπία ανάμεσα στην εξυγίανση και το δίκαιο περί των κρατών μελών. Και αυτή τη στιγμή ε, αναρωτιόμαστε αν... Ε, Άσχετα από τον λόγο της αφαιρεγγιότητας, ε, θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα καθεστώς ε, ε, για τους πιστωτές. Και να φροντίσουμε να υπάρχει συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών στην κρίσιμη αγορά της υποδομής. Όσον αφορά λοιπόν το δίκαιο αφαιρεγγιότητας των κρατών μελών, θεωρείται ότι η εξυγίανση είναι πάντα η καλύτερη λύση. Ε, έχετε ε, εμπειρία από την ε, υπόθεση της Banco Popular, δεν μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε εκεί την εξυγίανση. Μήπως μπορείτε να μας αναπτύξετε ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα της εξυγίανσης σε σχέση με τις κανονικές διαδικασίες αφαιρεγγιότητας των κρατών μελών. Και επίσης να μας πείτε ποιες είναι οι συνέπειες για, την, ε, για τις υποδομές της αγορές. Για παράδειγμα, εάν ε, χρησιμοποιεί κανείς ε, το νόμο περιφερειακότητας αντί για ε, την εξυγίανση, αυτό θα έχει συνέπεια στην αγορά. Ε, μεγάλη ερώτηση. Να ξεκινήσω από τα πλεονεκτήματα ε, της ε, σε σχέση με την αφαιρεγκαιότητα. Νομίζω το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει με την Τραπεζική Ένωση ε, έχουμε ένα σύστημα σε δύο βήματα. Έχουμε περίπου 4.000 τράπεζες στην Τραπεζική Ένωση και εποπτεία των μεγαλύτερων 125 γίνεται μέσω του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, ενώ για τις υπόλοιπες γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά την εποπτεία, ο Ντανιέλ Λουί λέει συνέχεια ότι πρέπει να εναρμονίσουμε τους κανόνες ώστε όλοι να παίζουμε με την ίδια παρτιτούρα. Και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για την εξυγίανση. Η εξυγίαση ε, θεωρούμε ότι είναι για, τις, για τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους. Και συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση στο, ταμείο, στο ενιαίο ταμείο ε, εξυγίανσης ως ιστατή ε, λύση ενώ ε, σε περίπτωση όπου οι τράπεζες δεν χρειάζεται να ε, τηρούν ε, τις υποχρεώσεις MRL, τις ελάχιστες απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων, μπορούν να μπουν σε κανονική διαδικασία αφαιρεγγιότητας. Αναλογικότητα μπορείτε να πείτε, αλλά έτσι ξεκινούν οι διαδικασίες αφαιρεγγιότητες, οι οποίες θα πρέπει να εναρμονιστούν. Όταν μιλάμε για CCP όμως μιλάμε για τελείως άλλο αριθμό ε, οργανισμών και μιλάμε για οργανισμούς για φορείς που συνδέονται με τις μεγάλες τράπεζες. Έτσι λοιπόν η χρεοκοπία ενός CCP θα έχει ε, αποτέλεσμα ντομινό στις ε, τράπεζες αυτές και αντιστρόφως. Τώρα το ένστικτό μου λέει ότι θα πρέπει να αναρωτηθείτε εάν θέλετε να δημιουργήσετε εθνικό σύστημα ή εάν για αυτόν τον ε, μικρό αριθμό, σε ακόμα μικρότερο αριθμό κρατών μελών, ε, θέλετε να επιλέξετε ευρωπαϊκή προσέγγιση. και να συνδέσετε το θέμα αυτό με την εποπτεία των τραπεζών. Θα ήμουν λοιπόν μάλλον υπέρ μια ευρωπαϊκή λύση. διότι είναι πολύ λίγοι οι CCP, οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι. Ελπίζω αυτό να απαντάει κάπως. Εγώ κοιτώ τον αριθμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Νομίζω πάντως ότι θα είχε νόημα να κάνουμε κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κυρία Σουίνμπεργκ. Όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, ε, ε, θα αρκεί ένα NCWO για ε, το θέμα της αφαιρεγγιότητας. Νομίζω ότι στην εξυγίανση σε σχέση με την κανονική αφαιρεγγιότητα απαλωτριώνουμε κάποια περιουσιακά στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην έχουμε διαφορετική μεταχείριση. Σε διεθνές επίπεδο είχαμε ε, εντατικές συζητήσεις για το θέμα αυτό και υπάρχουν εδώ κάποια προβλήματα, ε, διότι οι κεντρικοί αντισυλλαμβανόμενοι έχουν αντισυμβαλόμενοι έχουν δικούς τους κανόνες, ενώ με την ε, εξυγίανση είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι ε, ε, έχει προβλεφθεί μια λύση για το θέμα αυτό μέσα στο επόμενο δεκάμινο. Παρακαλώ. Ο κύριος Τρεμόζα, κυρία Κόνικ, σας καλωσορίζω στο Κοινοβούλιο. Μέσα στον τελευταίο μήνα είδαμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις με διαφορετική αντιμετώπιση από πλευρά του SRB. Το Banco Popular θεωρήθηκε ότι μπορούσε να διασωθεί σύμφωνα με τους ε, κανόνε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Μπάνκα Τιβιτσένσε και η Μπάνκα Βένετα θεωρήθηκαν πολύ μικρές, ε, μη συστημικές και έτσι εφαρμόστηκε το Ιταλικό Δίκαιο. Τελικά τα χρήματα του Ιταλού φορολογούμενου χρησιμοποιήθηκαν ε, πριν την πώλησή τους στην τράπεζα Σαβάλλο, παρότι και οι δύο τράπεζες ήθελαν να συγχωνευτούν και να δημιουργήσουν μία τράπεζα με ε, ε, στοιχεία του ενεργητικού 60 δισεκατομμύρια. Στην περίπτωση της Banco Popular, το SRB έχει πληροφορίες σχετικά με τις εκροές κεφαλαίων πριν την εξυγίανσή της. Ε, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία που έχουμε από τι ε, Ισπανικές Αρχές και για τις Ιταλικές Τράπεζες. Δεδομένου ότι ήθελαν να συγχωνευτούν η αντιμετώπιση τους σύμφωνα με το Ιταλικό Δίκαιο σημαίνει ότι όλες οι τράπεζες κάτω των 60 ε, δισεκατομμυρίων θα βρίσκονται εκτός της εντολής του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, τη διαφορά ανάμεσα ε, στην Banco Popular και την Veneto και Vicenza. Η βασική διαφορά που διαπιστώσαμε ήταν ότι η Banco Popular με 150 δισεκατομμύρια ισολογισμό ε, είχε δανείσει πολλά χρήματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ε, θεωρήσαμε λοιπόν ε, ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να εξηγιανθεί. Και έτσι βολήθηκε η τράπεζα στη Σανταντέρ. Στην περίπτωση των δύο τραπεζών της Βενετίας, που επί αρκετό καιρό βρίσκονταν σε προβληματικά ύδατα, Πράγματι ήθελαν να συγχωνευτούν. Το αν όμω ε, αυτή θα ήταν μια βιώσιμη λύση ή όχι είναι κάτι που θα πρέπει να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τουλάχιστον ε, θα ήταν βιώσιμη λύση αν υπήρχε σημαντική αύξηση κεφαλαίου. Δεν μπορούσαμε λοιπόν εμεί να το αποφασίσουμε αυτό. Εμείς ε, πέρσι στον προγραμματισμό ε, εξυγίανσης ε, είχαμε ασχοληθεί και με τις τράπεζες αυτές. Όταν ενεπλάκημενο όμως ήταν αρκετά σαφές ότι δεν υπήρχε πρόσφορη κάποια ιδιωτική λύση και γι' αυτό καταλήξαμε ότι λόγω του τεράστιου βαθμού μόχλευσης ουσιαστικά είχαν χάσει σημαντικό μέρος των πελατών τους μέσα στο τελευταίο 24 μήνο και κρίσιμες λειτουργίες των τραπεζών αυτών μπορούσαν εύκολα να αντικατασταθούν από άλλους παράγοντες και έτσι δεν υπήρχε μεγάλη διασύνδεση. Και αυτά είναι τα δύο βασικά κριτήρια για τον καθορισμό του δημοσίου συμφέροντος. Θα ήθελα να διασκεδάσω το επιχείρημα ότι αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες με ισολογισμό λιγότερο από 75-60 δισεκατομμύρια δεν μπορούν ε, να διασωθούν. Πρόκειται για κριτήρια που εξετάζονται για την κάθε τράπεζα συγκεκριμένα. Και όπως είπα, θα μπορούσε να έχει ληφθεί τελείως διαφορετική απόφαση πριν από ένα-ενάμιση χρόνο. Οι τράπεζες αυτές είχαν τότε βαθμό μόχλευσης ώστε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε νόημα να περάσουμε σε εξυγίανση. Ελπίζω να απάντησε. Έχω ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Δεν ε, μου απαντήσατε σχετικά με την Banco Popular. Ε, δεν ήθελα εσκεμένα να παραλείψω την ε, απάντηση αυτή. Μας ενημέρωσαν ότι η τράπεζα είχε αντιμετωπίσει σημαντικό όγκο εκροών ρευστότητας. Εμείς δεν εξετάσαμε ποιος απέσυρε ε, κεφάλαια από την τράπεζα. Δεν είναι δικιά μας δουλειά, δεν μπορώ να απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση αυτή. Σαφές όμως ήταν ε, ότι κατά την παρακολούθηση της τράπεζά μας, την τρίτη που αποφασίστηκε ότι η τράπεζα αυτή είναι αφαιρέγγια, το ερώτημα ήταν εάν θα μπορούσε να έχει η τράπεζα αυτή αρκετή ρευστότητα για την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Παλώμα Λόπες, παρακαλώ. Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστούμε που ήρθατε να μας δείτε σήμερα. Για πέστε μας για την εξυγίανση και διάσωση της Banco Popular. Θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία η ταχύτητα της ε, παρέμβασης έγινε στο πλαίσιο της αγοράς. Τελικά όμως κατέληξε σε σπαζογεφαλιά. Η θυμιστική Ευρωπαϊκή Αρχή με αυτά που έκανε έχει αφήσει να εκκρεμούν πάρα πολλές αμφιβολίες και να πλανώνται πολλές σκιές. Εσείς μας λέτε ότι όλα γίνανε όπως πρέπει, όλα γίνανε πάρα πολύ ε, συντονισμένα και τελικά οι μέτοχοι και οι αποταμιευτές τα χάσανε όλα και γι' αυτό και σας λέω ότι το Συμβούλιο Εξυγένσης στην καλύτερη περίπτωση ήταν αμελές. Χρησιμοποιήθηκαν όλα τα κριτήρια που έπρεπε για τη διάσωση της τράπεζας. Γιατί άλλοι είχαν άλλου είδου αξιολόγηση και οι άλλοι ήταν ε, ανεξάρτητοι φορείς και λάβανε υπόψη τα στρες τεστ. Άρα, τελικά όσο έκανε το Συμβούλιο επιτάχυνε την κρίση της ρευστότητα. Και έτσι φτάσαμε στην μέρα της 5ης ε, Ιουνίου. Και ε, πέστε μας πώς το Reuters ανακατεύτηκε στη διαπίστωση της ε, προβληματικής κατάστασης τράπεζας. Κόνιχ, να σας απαντήσω. Μισό το έσβησε το μικρόφωνο κατά λάθο. Νομίζω ότι η διάσωση της Banco Popular στα πλαίσια της σχετικής οδηγίας ήταν μια κίνηση επιτυχής. Εξασφαλίσαμε να μην υπάρχει μεταδοτικότητα, επιμόλυνση και διατάραξη της ε, σταθερότητας της αγοράς. Κανένας δεν χαίρεται από διάσωση και από εξήγηση. Όμως οι μέτοχοι και αυτοί που δεν είχαν προνομιούχες μετοχές χάσανε τις τοποθετήσεις επενδύσεις τους, αλλά όταν οργανώνεται μια τέτοια διαδικασία πώλησης πρέπει κανείς να στοχεύει στο μικρότερο κακό και αυτό και κάναμε και εμείς Τώρα, μας είπατε την, για την αξιολόγηση της Deloitte σε σχέση με τα stress tests. Αυτή η αξιολόγηση της Deloitte ήταν κάτι το οποίο επιτάσσει ο κανονισμός. Θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση, θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητη αξιολόγηση. Θα πρέπει να ξέρει μέσω αυτής της αξιολόγησης η αρμόδια αρχή για το τι συνήθειες υπάρχουν και τι εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν. Το stress test είναι κάτι όλος διαφορετικό. Έγινε το 2014 και το 2016 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για κάποια σενάρια μελλοντικά, Άρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ σταματώ τώρα ε, την κρίση της εκροής του, της ρευστότητας την προκάλεσε με συνεργειές του το Συμβούλιο Εξυγένσης. Ε, δεν νομίζω. Το διαπιστώσαμε ότι κάτι συμβαίνει και κάποια στιγμή αναλάβαμε δράση όσον αφορά την απόφαση της ε, Κεντρικής Τράπεζας να κηρύξει την Τράπεζα αφαιρέγγια με επικείμενη τέλος πάντων αφαιρεγγιότητα. Δεν νομίζω ούτε ότι υπήρξε κάποια παραβίαση του απορρίτου. Πάντοτε αυτό το Συμβούλιο τα λαμβάνει ε, σοβαρά. Και σε μια συνέντευξη με είχε ρωτήσει το Bloomberg σχετικά και είπα ότι εξετάζουμε αυτή την τράπεζα που εξετάζουμε όλες τις τράπεζες. Αυτή είναι η μόνη φράση που είπα. Το Reuters είχε ένα δημοψήφισμα και αν θέλετε να βρείτε ποιος τους τα είπε ψάξτε αλλού, όχι σε σχέση με εμένα Επερώτηση. Θα είμαι πάρα πάρα πολύ σύντομη. Δύο δευτερόλεπτα ερωτησούλα. Και ποιος θα αναλάβει το κόστος ε, της ζημίας που υπέστησαν οι αποταμιευτές. Και Δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά δεν είχε επιπτώσεις η διάσωση σε προνομίους ομολογίχους ή καταθέτες. Όλα αυτά τα κάλυψε η τράπεζα που αγόρασε την Banco Popular και όλα είναι όπως πριν. Ευχαριστούμε κυρία Κένιχ που ήρθατε, λέει ο κύριος Ουρτάσον. Εγώ θέλω να εμείνω στο θέμα της διαρροής προς το Reuters. Εσείς αρνείστε τη διαρροή. Όμως ισχύει ότι πολλοί παρατηρητές θεωρούν ότι εκεί είναι η ρίζα του κακού σε σχέση με το πρόβλημα της ε, ρευστότητας. Για πέστε μας, κάνατε εσείς στο Συμβούλιο κάποια έρευνα στο ιστορικό της υπηρεσίας γιατί είναι σημαντικό αυτό για την τράπεζα. Θα ήταν σοφό να κάνετε τέτοια έρευνα για την έκθεση τώρα της Deloitte. Όντως αυτό το επιτάσσει ο κανισμός. Και μάθαμε ότι υπήρχαν τρία σενάρια σε εκείνη την αξιολόγηση. Το καλύτερο σενάριο, πέστε μου αν ισχύει κάτι τέτοιο, έλεγε για 1,5 δις αξιολόγηση. Το επιβεβαιώνεται Επίσης, ποια είναι τα κριτήρια του Συμβουλίου Εξυγένσης. Πώς αποφασίζετε ποια αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη. Τι κριτήρια έχετε. Και επίσης πάλι για την Deloitte. Για μου το Συμβούλιο προτίθεται να δημοσιοποιήσει αυτή την αξιολόγηση ή υπάρχει ε, κάτι, κάποια διάταξη που το απαγορεύει. Και τελευταία ερώτηση. Τι γίνεται με τον αντιπρόεδρο της Τράπεζας της Ισπανίας που έλεγε ότι υπήρχαν και άλλα στοιχεία εγγύησης στην τράπεζα με τα οποία θα μπορούσε η τράπεζα να πάει στα πρότυπα τλάκ. Είχαν ισχύει κάτι τέτοιο. Για να τα αρχίσω από το τέλος, λέει η, η κυρία Κένιχ το σχόλιο που έγινε από τον υποδικητή της Τράπεζας Ισπανίας πρέπει να μιλήσετε μαζί του. Εμείς ενημερωμήθηκαμε την Τρίτη το βράδυ ότι αυτή η τράπεζα δεν ήταν σε θέση να καλύψει το έλλειμμα ρευστότητας. Και ε, ε, δεν έκλεισε η τράπεζα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ε, σχετικά με την έκθεση Deloitte για την ώρα δεν υπάρχει πρόθεση δημοσιοποίησης της έκθεσης, περιέχει πάρα πολλές εμπιστευτικές ε, πληροφορίες, αλλά υπάρχουν Υπάρχουν δύο εκθέσεις για την ώρα. Μία αξιολόγηση της λογιστικής κατάστασης της τράπεζας και η δεύτερη κατάσταση είναι η ανεξάρτητη αξιολόγηση που θα γίνει από μια εταιρεία λογιστική, από κάποιον αρμόδιο φορέα που ε, να ε, πληροφορεί τις ε, αρχές εξυγίανσης για τις οικονομικές επιπτώσεις των διαφόρων εργαλείων. Δεν μπορώ να πω ότι κάναμε σήμερα, μας χρειάστηκε χρόνος. Έχουμε δημοσιοποιήσει σήμερα ε, μια εκδοχή της απόφασης εξηγίασης που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας που περιέχει όλες αυτές τις ε, πληροφορίες που δεν ε, θεωρούμε ευαίσθητες από την άποψη της εμπιστευτικότητας και, και εσωτερικά έρευνα βεβαίως, η, για μένα η απάντηση είναι πάρα πολύ ε, εύκολη, ε, δεν ήταν όμως εύκολη για όλη την Ευρώπη. Διάβασα ε, με κάποια καθυστέρηση διότι βρισκόμουν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ναι, σχετικά με τα διάφορα σενάρια της έκθεσης Deloitte. Υπήρχαν τρία σενάρια όπως γνωρίζετε. Τι πιο ε, ποιο χρησιμοποιήσατε θετικό ή αρνητικό σενάριο, διότι αυτό κάνει τη διαφορά. Ναι, χρησιμοποίησαμε το, το δύο στην έκθεση για να ε, τεκμηριώσουμε την απόφασή μας αλλά χρειάζεται κανείς ε, μια, έναν αγοραστή και την τιμή που προσφέρει ο αγοραστής σε μια τέτοια περίπτωση. Ευχαριστώ. Μπάρμπαρα Κάμπελ. Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Κιόνικ που βρίσκεστε δεύτερη φορά εδώ στην Επιτροπή μας. Επιτρέψτε μου μία ερώτηση σχετικά με το ερώτημα εξυγίανση σε σχέση με την αφαιρικαιότητα. Δεν ξέρω να έχω καταλάβει σωστά. Είδαμε στην Ιταλία τις δύο τράπεζες, την Βενέτο και την Ποπολάρη τη Βιτσέντσα, ε, να περνάνε από την εθνική διαδικασία αφαιρικαιότητας. Ε, και είπατε ότι ε, σε ιδανική περίπτωση θα έπρεπε να, εναρμονιστεί, να εναρμονιστούν τα εθνικά δίκαια αφαιρεγγιότητας. Ε, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν σήμερα είδαμε τη διαδικασία εξυγίανσης. Ε, και άλλη ερώτηση. Είπατε ότι στο SRF έχουν 6,6 δισεκατομμύρια έχει δώσει κάθε κράτος ε, για το ε, Ταμείο Εξυγίανσης. Ε, μπορείτε να μας μιλήσετε σχετικά με αυτό και όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικά τα σχέδια εξυγίανσης για να αποφασίσουμε αν θέλουμε προσέγγιση ενιαίου ή πολλαπλών σημείων εισόδου. είναι σημαντικό να ληφθεί σχετική απόφαση, διότι οι δύο προσεγγίσεις έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το single point of entry μάλλον είναι καλύτερο ε, για τράπεζες ε, στο ίδιο στην ίδια δικαιοδοσία, ενώ το multiple point of entry μάλλον είναι πιο χρήσιμο για διάφορες ε, άλλες ε, σκόρπιες τράπεζες και υπάρχει και η μεικτή λύση. Εσύ σε ποια λύση θεωρείτε πιο ιδανική. Καταρχάς όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση. Α, όχι, θα το πω αγγλικά. Αν κατάλαβα απόλυτα καλά, έχουμε σύστημα ώστε να έχουμε για τις μικρές τράπεζες αφαιρεγγιότητα, διαδικασία αφαιρεγγιότητας ε, και μόνο για μεγάλες τράπεζες δημοσίου συμφέροντος ε, για τα κράτη-μέλη και για την Ένωση στο σύνολό της ε, θα προβλέπεται η διαδικασία εξυγήνσης, το οποίο σημαίνει ότι και για τις μικρές τράπεζες δεν θα, θα χρειαστεί να εκπονηθούν σχέδια εξυγίανσης, δεν θα υπάρχουν ε, απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων, όμοιες με αυτές ε, των μεγάλων τραπεζών. Μόνο λοιπόν για τις πολύ μεγάλες τράπεζες θα πρέπει να καθοριστούν τα MRL ε, και να υπάρχουν σχέδια εξυγίανσης. Όσον αφορά το ε, ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, όλα προχώρησαν σύμφωνα με τα σχέδια μας. Εδώ στις Βρυξέλλες κάναμε τους υπολογισμούς μας και τα κράτη-μέλη συνέλεξαν τους πόρους και τους μετέφεραν νομίζω τώρα στις 30 Ιουνίου νομίζω ήταν η προθεσμία. Τα πράγματα αυτά λοιπόν ε, προχωρούν σωστά. Εξυγίανση και ενιαίο ή πολλαπλά σημεία εισόδου. Ποια είναι η δική μας προτινόμενη στρατηγική. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε ε, ε, ε, στρατηγική που να προτιμούμε, διότι όλα εξαρτώνται από την οργάνωση της ίδιας της τράπεζας. Αν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός, αν η χρηματοδότηση είναι, γίνεται κεντρικά στο πλαίσιο της τράπεζας, τότε το single point of entry μάλλον είναι ο η σωστή στρατηγική. Αλλά και τα πολλαπλά σημεία εισόδου μπορεί επίσης να είναι κατάλληλη στρατηγική για τράπεζες που έχουν ανεξάρτητες θεατρι... Και νομίζω ότι στη συνέχεια θα δούμε πολλές ενδιάμεσες περιπτώσεις. Δηλαδή να έχουμε ενιαίο σημείο εισόδου για κάποιες τράπεζες ε, με θηγατρικές σχετικά ανεξάρτητες ε, που ενδεχομένως να εξεταστούν ξεχωριστά ή να έχουμε και περιφερειακούς κόμβους. Ε, πάντως ε, δεν μπορείτε να επιλέξετε εσείς ποιο μοντέλο προτιμάτε. Ε, τα συστήματα αυτά ακολουθούν τον τρόπο οργάνωσης της τράπεζας. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση, δηλαδή για λόγους διαχείρισης κινδύνου να έχουμε το, τα πολλαπλά σημεία εισόδου, τότε αυτό θα αντικατοπτρίζεται στον σχεδιασμό για, τις, ε, για την εξυγίανση. Ε, ο πρόεδρος Διακόπτη έχει λήξει ο χρόνος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Έχω δύο ή τρεις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, πώς εξηγείται το γεγονός ότι η Banco Popular τον Ιούνιο 2016 έκανε ανακεφαλαιοποίηση 2,5 δισεκατομμυρίων και μεταπτώχευσε τον Ιούνιο του 2017 παρά το γεγονός ότι το δυσμενές στενάριο των stress test για, να, για τις κεφαλαίων της ε, τράπεζας δεν ε, υλοποιήθηκε όσον αφορά την ισπανική οικονομία. Αντίθετα, η ισπανική οικονομία, κατά την άποψή μου, βαίνει καλώς. Δεύτερη ερώτηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, μου φαίνεται ότι η εξυγίανση της Banco Popular υλοποιήθηκε με τρόπο ώστε δεν κόστισε τίποτα ε, στο Συμβούλιο Εξυγίανσης, στο ΕΝΙΑ, και δεν κόστισε τίποτα ε, στην, ε, στο κράτος, στο Ισπανικό και στον φορολογούμενο τον Ισπανό. Αυτή είναι η περίπτωση πράγματι, διότι αν είναι αυτή η περίπτωση θα πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία αυτή η εξηγήση, αλλά υπάρχουν ίσως μερικές έμμεσες, έμμεσο κόστος που δεν κατανόησα που δεν αντελήφθην. Και τρίτη ε, ε, ερώτηση, ε, σύμφωνα με τον ΕΡΙΑ, για την Τράπεζα Βένετο, δύο ορισμοί χρησιμοποιήθηκαν, ένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας άλλος σε επίπεδο εθνικό. Μου φαίνεται ότι η διαφορά ίσως υπομονεύει την συνεκτική εφαρμογή ε, του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την εξυγίανση. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Το ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν μπορώ να σχολιάσω το γεγονός ότι το 2016 ε, έκανε ανακεφαλοποίηση και το πτώχευσε το 2017. Το 2017 η δίκηση της τράπεζας αναγνώρισε ότι ε, χρειαζόταν μια ε, καθάριση κατά κάποιο τρόπο, μια, να βάλει τάξη και να λάβει υπόψη τις ζημίες. Αλλά αυτό είναι θέμα εποπτείας, δεν είναι δικό μας θέμα. Το γεγονός ότι τα stress test ε, δεν αποκαλύψαν την κατάσταση έδειξαν ότι στο δυσμενές σενάριο ήταν η τράπεζα ε, μεταξύ ε, που είχε το μεγαλύτερο χάσμα, τη μεγαλύτερη διαφορά με τη γραμμή βάσης, αλλά και αυτό είναι θέμα εποπτείας, ε, κόστος για τον φορολογούμενο, κόστος για τρίτα μέρη, όχι δεν νομίζω, είπα και προηγουμένως ότι πουλήθηκε η τράπεζα στην Σανταντέρ χωρίς ε, καμία ρεσιμότητα, χωρίς όρους. Η Σανταντέρ είναι ο ιδιοκτήτης δεν υπήρξε κανένα κόστος για το φορολογούμενο, κανένα κόστος για άλλες, άλλους φορείς και ήταν μια τράπεζα όπου μπορούσαμε να προστατεύσουμε τους ομολιούχους υψηλής εξασφάλισης και η τράπεζα και τα υποκαταστήματά της άνοιξαν την επόμενη μέρα σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Ο Ανδρεανδρίας είδα τη δήλωση για την Βένετο ε, το θέμα ήταν διαφορετικό από ευρωπαϊκής ε, και από εθνικής απόψεως είπατε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο κρίσιμο αυτό. Εξετάσαμε το δημόσιο συμφέρον με την έννοια ε, της οδηγίας πρόκειται για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η Ιταλική κυβέρνηση εξέτασε πολύ περισσότερα θέματα απασχόλησης, κοινωνικά θέματα και ε, είχε μια μικρο άποψη του αντικτύπου. Αλλά αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί από τις εθνικές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου Εξυγένσης. Νομίζω ότι η διάσωση της Banco Popular ε, χαρακτηρίζεται από κάποιες σκιές που θα πρέπει να τις φωτίσουμε. Τώρα είμαστε στην πρώτη φάση και νομίζω ότι το Συμβούλιο Εξηγένσης επέδειξε κάποια μη συνετή στάση. Στη συνέχεια δε υπήρξε άρνηση για οποιοδήποτε σχόλιο. Όχι, δεν λέω ότι σε δική σα δηλώση οφείλεται η διαρροή προ το Reuters και ούτε οφείλεται σε κάποιο μέλο του Συμβουλίου. Από την άλλη μεριά όμω, ε, το ότι κατονομάσατε μια συγκεκριμένη τράπεζα στο Bloomberg, ε, αυτό ήταν τουλάχιστον ε, άφρον, ασύνετο. Οπότε δεν λέω, ότι οι δηλώσεις έφεραν την νεκροή των κεφαλαίων, αλλά ε, έβαλαν ένα χεράκι. Το θέμα είναι εσείς στο μέλλον θα κατονομάζετε τράπεζες που είναι στη φάση της εξέτασης από το Συμβούλιο Εξυγένσης. Κατόπιν αυτής της φάσης των δημοσίων δηλώσεων υπήρξε η φάση που ήταν η τέλεια σιωπή από πλευρά του Συμβουλίου. Εντάξει, η έκθεση Deloitte ήταν ε, ε, εμπιστευτικού χαρακτήρα. Τι γίνεται όμως με την εκ των υστέρων ανάλυση που στο ε, άρθρο 20 στο σημείο 16 προβλέπει ο κανονισμός δεν θα πρέπει να αναλυθεί το πώς αξιολογήθηκε η απόφαση ή τέλο πάντων η κατάσταση για να λυθεί η απόφαση. Και σήμερα το πρωί ο κύριος Ντομπρόφσκης, ο Επίτροπος, είπε ότι είναι αγώγιμη αυτή η απόφαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχει δηλαδή ένδικο μέσο για να προσφύγει κανείς εκεί κατά της απόφασης. Νομίζω ότι θα πρέπει στην φάση της ανάλυσης να υπάρχει απόρριτο από πλευράς υποπτίας, αλλά αφού αναλυθούν ενέργειες θα πρέπει να υπάρχει τέλεια διαφάνεια. Εγώ νομίζω ότι το αντίθετο έγινε, το, το αντίστροφο όσον αφορά την περίπτωση Banco Popular. κυρία Κένιχη. Κατηγορηματικά θα απαντήσω αρνητικά στο ότι είχα αμετροέπεια όσον αφορά ε, τις δηλώσεις. Να κάνουμε πίσω να τα δούμε ε, πάλι. Ποτέ στο Συμβούλιο δεν ε, σχολιάζουμε συγκεκριμένες τράπεζες. Το σχόλιο στο οποίο προέβην είναι το μόνο το οποίο βέβαια έδειξε τηλεόραση το ότι με ρώτησαν, ε, με ρώτησαν το ε, εάν εξετάζουμε αυτή την τράπεζα και είπα ότι την εξετάζουμε αυτή την τράπεζα όπως και άλλες πολλές τράπεζες. Αυτό θα μπορούσα να το πω για όλες τις τράπεζες και το έχω πει πολλές φορές για όποτε με ρώτησαν για το τι κάνουμε. Μα αυτή είναι η δουλειά μας, εξετάζουμε τις τράπεζες. Και όσον αφορά το Reuters, όπως προείπα, είναι άλλο θέμα. Ρωτήστε το Reuters α, ποια ήταν η πηγή του. Δεν ήμουν εγώ πάντως. Τώρα όσον αφορά την σιγή που ακολούθησε, αυτό επιτάσσεται από τον νόμο. Από το πρωί δηλαδή της 7ης Ιουνίου. Οπότε και σωστά δημοσιεύσαμε μια σύνοψη της αποφάσεως εξηγήνσης. Γιατί ο νόμος επιτάσσει είτε να υπάρχει αυτή η δημοσίευση της σύνοψης, είτε να υπάρχει ε, δημοσίευση της πλήρους αποφασίσεως αποφάσεως συγγνώμη, με την διαγραφή οποιοδήποτε στοιχείου διαβαθμισμένου και απορρίτου. Επειδή όμω αυτό θα κάνουμε 7 η ώρα το, το, πρωί, ε, κάναμε ότι ήταν πιο εύκολο, πιο σύντομο. Αν αυτό γινόταν σήμερα, Οπότε και γι' αυτό και δημοσιεύσαμε την ε, απόφαση αφαιρώντας Αυτά τα οποία κρατήσαμε με το κοινοτικό δίκαιο ήταν ε, εμπιστευτικού χαρακτήρα. Τώρα. Για να διασαφίσω την επόμενη ερώτηση. Ε, βέβαια και χρειάζεται διαφάνεια και φροντίζουμε να υπάρχει. Έχει δίκιο ο κύριος Ντομπρόφης, γι' αυτό εννοούσε. Όποιος θεωρεί ότι έχει φυγεί από τις ενέργειές μας έχει δύο λύσεις. Πρώτα πρώτα να προσφύγει στη διοικητική δικαιοσύνη. Τώρα δεν ξέρω έτσι, νομίζω, δεν, δεν είμαι νομικός. Άλλη λύση είναι να προσφύγει κανείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Συνεργές μας, μια που λάβαμε αυτή την απόφαση της διάσωσης και την εφήρμαση την απόφαση μας το Ισπανικό κράτος. Και να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Προσπαθούμε να λάβουμε την ορθότερη δυνατή απόφαση. Εποφελία της ε, σταθερότητας της ε, σπανικής οικονομίας, των ε, μετόχων και των καταθετών. Θα γίνει μια εξπόστ αξιολόγηση. Ναι, ναι, ναι, την προετοιμάζουμε. Είναι το επόμενο βήμα. Ο κύριος Μάτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μας μιλήσατε για τον Κοκοκουλάρη, μας μιλήσατε για τις τελικές τράπεζες και συμφωνώ ότι ικανοποιητικά πήγαν τα πράγματα στον αφορά την Ισπανική Τράπεζα. Αλλά συμφωνείτε ότι είναι κάπως παράδοξο ότι είναι δυνατόν να εγκριθούν κρατικές ενισχύσεις ε, όταν υπάρχει κάποια απειλή διατάραξη όταν το Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να ξεκινήσει διάσωση γιατί δεν υπάρχει ε, γενικό δημόσιο συμφέρον προς τούτο. Επίσης, έχω και μια άλλη διαφορετική ερώτηση όσον αφορά το Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων. Αυτό μας καίει όλους, γιατί υπάρχει μια απόφαση, μια πρόταση που θα κλείσει δύο χρόνια. Και τι γίνεται όσον αφορά ε, αυτού του είδους την, την πάρα πολύ βραδία πρόοδο Οπότε θα ήθελα να μου πείτε την ε, γνώμη σας. Θεωρείτε ότι στα πλαίσια όλων αυτών των θεμάτων που εκκρεμούν έχουμε και τις ε, εκλογές που έρχονται, έχουμε την ατμόσφαιρα και ίσως γι' αυτό το λόγο δεν έχει προοδεύσει αυτή η υπόθεση, αυτό το ντοσχεία. Τι λέτε εσείς όσον αφορά αυτή την έλλειψη πρόοδου θεωρείτε ότι θα υπάρξει αλλαγή στάση από πλευρά τη Επιτροπή, ούτω ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα. Κιόνι. Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση του γιατί δόθηκαν οι κρατικές ενισχύσεις ε, σε μια περίπτωση κατά την οποία εμείς είπαμε ότι δεν υπάρχει δημόσιο συμφέρον για διάσωση η ερώτηση θα πρέπει να απευθύνει σε αυτούς που έλαβαν την απόφαση Ιταλική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή. Αλλά να σας πω περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω ότι επρόκειτο για ενίσχυση όσον αφορά ε, την ρευστότητα. Το είπε ο Πρόεδρος. Πάντοτε χρειάζεται κάποιο είδου ε, περιθώριο λιγμών, ακόμα και σε περίπτωση εκαθάριση, για να βοηθηθεί η εκαθάριση. Τώρα για τις λεπτομέρειες ας είμαστε προσεκτικοί. Τέτοιου είδου ενισχύσεις πάνε και σε άλλους κλάδους. Πάντως η τραπεζική εξηγήνση πάντοτε θα πρέπει να συνοδεύεται από την ελάχιστη δυνατή συνέπεια για τους ε, καταθέτες. Και εμείς όπως και εσείς έχουμε την ίδια φιλοδοξία να θεσπιστεί σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Ένα σύστημα που τέτοιου είδους ασφάλισης, αντασφάλισης αρκεί σήμερα, δεν ξέρω, συζητήσιμο, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινή εποπτεία κοινό καθεστώς διάσωσης. Όμως, αν κάτι πάει στραβά, τι γίνεται. Τότε τι θα κινδύνο τα εθνικά συστήματα ε, εγγύησης των καταθέσεων. Πολλά, πολλά ε, βρίσκονται στο τραπέζι για συζήτηση. Όχι, δεν θα κρεμούν για πολύ όμως. Ευχαριστώ πολύ ο Γιάκοπ ε, κυρία ε, δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη έχει να κάνει με τη δυνατότητα διάσωσης ε, προνομιούχων μετοχών, ε, ομολόγων. Συγγνώμη φαίνεται να ε, αρχίζει να υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την διάσωση των ομολόγων αυτών. Ε, σχετικά με το αν θα γίνει στην πράξη, δηλαδή, παρότι θεωρητικά ε, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διάσωση. Και το θέμα είναι αν η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού επιτρέψει λύση για κάποια από τα θέματα που αναφέρατε και το γεγονός ότι δεν συμπεριέλαβε την διάσωση των ομολόγων, διότι θεωρήθηκε μη βιώσιμη λύση. Ταυτόχρονα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το MRL και το TILAC, τη δυνατότητα απορρόφησης βασίζεται στην προϋπόθεση ότι μπορούν και στην πράξη να ε, αποτελέσουν αντικείμενο διάσωσης ε, οι ε, τα ομόλογα αυτά. Η δική σας θέση ποια είναι θα μπορέσει να γίνει αυτό. Είναι σωστή η η υπόθεση αυτή των αγορών και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο όταν εξετάσουμε την νομοθεσία ε, σχετικά με το MRL και το TILAC. Το άλλο θέμα είναι αυτό που έχει να κάνει με το κεντρικό αντισυμβαλόμενο. Ε, εδώ μπορεί να υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε ε, να έχουμε και για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους αυτό που έχουμε για, την, για τις τράπεζες, δηλαδή έναν ενιαίο επόπτη. Αυτό όμως θα οδηγήσει και στο ερώτημα εάν θα πρέπει να υπάρχει και μία ενιαία αρχή ε, για την ε, ανάκτηση και εξυγίανση. Και αυτό οδηγεί με τη σειρά του στο ερώτημα αν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό μέσο στήριξης ε, ή εξυγένσης. Πώς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να οργανωθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ να προσπαθήσω να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Νομίζω ότι, ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες, πρέπει να είμαστε όμως απόλυτα σαφείς. Η οδηγία για την ανάκαψη και την εξυγίανση δεν αποκλείει αυτά τα ομόλογα από τη διάσωση και αυτό για μένα θα ήταν και λάθος μήνυμα, ε, διότι πρόκειται για μέσο με ε, πιστοτικό κίνδυνο και γι' αυτό στην ιεράρχηση ε, θα πρέπει να μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διάσωση και στις τράπεζες όπως και σε, οποιαδήποτε άλλη, σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Σχετικά με το αν αυτό είναι πολιτικά βιώσιμο ή όχι, θα πρέπει να εξετάσει κανείς ε, την κατάσταση του συστήματος σε σήμερα. Ήδη έχει κληρονομήσει κάποια τέτοια θέματα και ε, ο ε, κάτοχος των, κρατικών, ομολόγων αυτών είναι πελάτης της τράπεζας. Εάν λοιπόν Ε, προχωρήσουμε σε εξυγίανση των πελατών, αυτό που αφήνει την τράπεζα. Ε, εσείς το συνδέετε αυτό και με τη δέσμη μέτρων για τον MRL. Τις ελάχιστες απαιτήσει ε, ιδίων κεφαλαίων, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση και να φροντίσουμε να υπάρχει κεφάλαιο που να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διάσωσης. Δεν ε, θα έλεγα όμως ότι όσοι κατέχουν ε, τέτοια ομόλογα είναι ε, πάντα ασφαλείς. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι σαφές. τα ομόλογα αυτά αποτελούν πιστοτικό μέσο σε οποιονδήποτε τομέα. Και στην άλλη ερώτηση νομίζω ότι απάντησα εν μέρη όταν απαντούσα στην κυρία Σουίνμπερν. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε για το σχετικά μικρό αριθμό κεντρικών αντισυμβαλωμένων ε, να έχουμε μία ενιαία αρχή ε, η οποία να συνδέεται και με, την, ε, με τις τράπεζες, διότι υπάρχουν εδώ πολλές αλληλεξαρτήσεις. Σχετικά με το αν χρειαζόμαστε ταμείο εξυγίανση. Εγώ θα έκανα ένα βήμα πίσω και θα εξέταζα ε, ποιο είναι το απαραίτητο κεφάλαιο ε, για την εξυγίανση ενός κεντρικού αντισυμβαλωμένου. Η Ευρώπη δεν νομίζω ότι έχει δώσει ακόμα απάντηση στο θέμα αυτό. Και επειδή ασχολούμαι με το θέμα αυτό και σε παγκόσμιο επίπεδο, το θέμα αυτό έχει τεθεί στο θεματολόγιο τη επόμενη χρονιά. Να εξετάσουμε δηλαδή πόσο πρόσθετο κεφάλαιο να είναι απαραίτητο ε, και για να έχουμε και μέσω στήριξη, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια τη κυρία Περέ. Ε, φαίνεται λοιπόν ε, να υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε όμως να το ε, ποσοτικοποιήσουμε ακόμα. Και το TILAC και το MRL μάλλον δεν είναι η λύση για τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους. Ευχαριστώ πολύ. Προτείνω να συνδυάσουμε τις δύο τελευταίες ερωτήσεις Καστιάη. Ο κύριος πρώτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και κανείς δεν ξέρει πραγματικά εάν θα μπορέσουμε να τα μειώσουμε με τρόπο ε, αποτελεσματικό και ικανοποιητικό. Αν παραμείνουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο, αυτό θα έχει αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο. Πιστεύετε ότι η κατάσταση θα προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. περβάσου Μπέρες. Κυρία Κόνιγκ, αρχίσατε να μιλάτε για τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την πρώτη εφαρμογή ε, σημαντική των ε, εργαλείων της οδηγίας, αλλά δεν αναφέρατε για τον αντίκτυπο στην αγορά. Μήπως δεν υπάρχει θέμα σε αυτό το επίπεδο. Με, το οδηγία, με την οδηγία υπάρχει μια αναδιάρθρωση της αγοράς που οργανώνεται. Βεβαίως αυτό είναι πέραν ε, της δικής σας εντολής, αλλά παρόλα αυτά έχετε ένα παρατηρητήριο για να δείτε πώς ε, η οδηγία αυτή ε, εξυγίανσης ε, παρεμβαίνει στη λογική της αγοράς και στα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανταλλάσσονται με αυτές τις συνθήκες και μήπως ε, μια νομοθεσία που έχει προκυκλικό αντίκτυπο κυρίως όταν βλέπουμε ε, την ε, τιμή της μετοχής της Banco Popular και την προοπτική στη διάρκεια. Κύριος Καλβέ ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Είμαι, χαίρομαι πολύ ε, για την εξυγίανση της Banco Popular. Είμαι πελάτης της Banco Popular και για μια φορά ε, βεβαίως δεν πλήρωσαν καταρχήν οι φορολογούμενοι. Βεβαίως θα υπάρξουν απαιτήσει αγωγές ε, στην, ε, στο δικαστήριο, θα υπήρχαν ούτως ή άλλως. Έχω δύο ερωτήσεις σχετικά με τις ακτιβιστές στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Βεβαίως, η εξυγίανση ήταν καλή, αλλά δεν νομίζετε ότι πρέπει να δούμε τι συνέβη πριν από την εξυγίανση, η αναθεώρηση, ο έλεγχος, διότι ο κύριος Κωνστάνσιο μου είπε βεβαίως η, η ε, ε, εγκρίθηκε, ε, πρέπει όμως να επινοήσουμε κάτι. μου είπε πρέπει να ελεγχθεί. Τι πιστεύετε για το γεγονός ότι η Popular πηγαίνει Σανταντέρ, έχουμε τις Ιταλικές τράπεζες τώρα που de facto ε, ε, μικραίνει η Τραπεζική Ένωση, οι διασυνοριακές χάνουν δεκασεκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτές. Αυτές οι ερωτήσεις είναι περισσότερο για την εποπτεία. Τις καλύτερα να θεθούν στην εποπτεία. Θα ήθελα με αυτή τη σειρά να πω ότι συμφωνώ μαζί σας ότι σε αυτές τις δύο περιπτώσεις ότι ήταν μάλλον εθνικές λύσεις και όχι διασυνοριακές λύσεις ε, διευρωπαϊκές. Δεν είναι πάντοτε η περίπτωση. Είχαμε άλλες περιπτώσεις στην Πορτογαλία όπου τράπεζες ε, διασυνοριακές ε, από άλλη χώρα ανέλαβαν την κατάσταση. Ε, περνάμε σε ένα βεβαίως πιο διεθνές πλαίσιο. Η πρώτη ερώτηση βεβαίως είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από νομισματικής ε, πλευράς και από πλευράς εποπτείες ε, διδάγματα. Βεβαίως ότι οδηγεί η οδηγία αυτή σε αναδιάρθρωση της αγοράς. Συμφωνώ μαζί σας κυρία Πέρες ότι ελπίζω ότι η αγορά κατανοεί, κατανοεί και ότι πρέπει να αξιοποιήσει λογή το τίμημα ε, του κινδύνου. Ε, δεν υπάρχει ε, βεβαίως δωρεάν ανόρθωση και το κράτος να αναλαμβάνει τα πάντα. Η Banco Popular απέδειξε πολύ καλά και καλά αντέδρασε ορθολογικά η αγορά. Για την Ελλάδα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα και Κύπρο βρίσκονται τα κόκκινα δάνεια σε υψηλό επίπεδο πληροφορηθήκαμε από τον μηχανισμό, τον ενίο μηχανισμό εποπτείας ότι, ότι εργάζονται σκληρά για το θέμα αυτό των κόκκινων δανείων των τραπεζών. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά και η εργασία που γίνεται παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για τις, ε, τα θέματα σχετικά με τον νόμο αφαιρεγγιότητας και πτώχευσης ε, και θα μπορούσε να υπάρχει βεβαίως αυτό ένα, ε, ένα παράδειγμα, ένα, μια μέθοδος και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Βεβαίω και το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί ότι οι υποθέσεις αναδύονται, θα προβληματιζόμαστε, αλλά πάντως ευχαριστούμε για την προθυμία σας να τα συζητήσουμε. Και σημαντικό συμπέρασμα για το μέλλον είναι ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία και να έχουμε τα σχετικά μέσα στα μέτρα προστασίας, να βλέπουμε τα θέματα της ρευστότητα ε, και η στήριξη είναι σημαντική. Αλλά επίσης η εγγύηση για τις καταθέσεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αξιολόγηση των ισχυών των κανόνων. Είναι αυτό που λέγαμε. Διακοπή 30 λεπτών. Και θα συνεχίσουμε στις 6 με τον mm -hmm. Εστονό Υπουργό. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό Οικονομικών της Εστονίας και Πρόεδρο και Προεδρεύοντα σωστότερα του ΕΚΟΦΗΝ, τον κύριο Τόμας Τόνιστε. Σας ευχαριστούμε κύριε που απεδέχτετε την πρόσκλησή μας και ήρθατε για να συζητήσετε με την Οικονομική Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Και προσβλέπουμε στην συνεργασία με εσά, το επιτελείο σας και γενικότερα την ε, ε, Στονική Προεδρία. Ελπίζουμε σε μια εργαστή συνεργασία, ούτως ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Περιμένουμε τις προτεραιότητές σας και είμαι σίγουρο ότι θα είναι παραγωγική η συνεργασία μας. Έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να ζητηθούν στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και φυσικά μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων του επόμενου εξάμεινου. Θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα είναι αρμονική. Οπότε η Οικονομική Επιτροπή μας εύχεται καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ρομπέρτο, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Με τιμάει η πρόσκλησή σας και θα σας μιλήσω στα εστονικά. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε την υπέροχη γλώσσα μας. Έλεγα ότι με τιμά η πρόσκλησή σας και σας ευχαριστώ. Μου δίνει ευκαιρία να παρουσιάσω για τα οικονομικά και νομισματικά τις προτεραιότητες μας. Είναι συμβολικής μεγάλης σημασίας η άσκηση της Προεδρίας. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Και όπως η ομολογή μου Είμαι και εγώ βαθύτατα ευρωπαίος, πρόκειται για την ειρήνη, πρόκειται για την δημοκρατία και αυτά είναι και αξίες που και προσωπικά ενστερνίζομαι. Εκτιμώ πάρα πολύ τις ελευθερίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν κατοχήθει για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Ξέρω ότι θα πει να τα αποστερείτε κανείς. Ξέρουμε εμείς τι σημαίνει επομένω το να μην υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα. Σας διαβεβαιώ ότι η Προεδρία μας δεν θα έχει ως περιεχόμενο ε, όνειρα και οράματα. Να σας πω ποιες θα είναι τα δραστηριότητες που θα διατηρήσουν αυτή μας την ε, Προεδρία. Σε αυτή την συγκυρία η οικονομική ανάπτυξη συνεχίζει να ανεβαίνει. Έχει υποχωρήσει η αβεβαιότητα που προηγήθηκε και είναι ενθαρρυντικό το ότι η οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη δημιουργεί θέσεις εργασίας και μειώνονται οι άνεργοι. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να επαναπαυθούμε και να, ε, να στις δάφνες μας θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη θετική οικονομική συγκυρία, τις ευκαιρίες που προσφέρονται για να μπορέσουμε να πετύχουμε πρόοδο και να έχουμε καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ούτω ώστε να έχουμε μια μακρόπνοη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Όσον αφορά τον συντονισμό ε, και οικονομικής πολιτικής, θα πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας σε πιο σωστή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που φέρνουν την ε, ανάπτυξη. Να ακολουθήσουμε τις αναχώρα συγκεκριμένες συστάσεις. Ε, κλείσαμε ήδη μια συμφωνία όσον αφορά τους ε, στόχους για το 2018 όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και είπαμε ότι θα δούμε πώς θα έχουμε όσον αφορά περισσότερη ανάπτυξη με την εφαρμογή των συστάσεων. Αυτό θα γίνει με αμοιβαία υποστήριξη και επισημάνσεις. Να έχουμε μια δημοσιονομική πολιτική που να οδηγεί σε βιώσιμα δημοσιονομικά. Να βοηθούνται έτσι οι οικονομίες. Η Προεδρία πρέπει να διασφαλίζει την ταχεία λήψη αποφάσεων που βοηθούν στο Συμβούλιο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για αποφάσεις που θα υποβληθούν τους αμέσως επόμενους μήνες στο Συμβούλιο. Θέλουμε διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις και αυτό σαφώς είναι κάτι που να κάνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχουμε έμεσες συνέπειες θετικές στην ε, Ευρωζώνη. Όσον αφορά το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, έχουμε ακόμα κάποιες ε, αντιθέσεις μεταξύ των εθνικών πολιτικών και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ας πούμε, είναι κάτι το οποίο πρόσφατα τονίστηκε ε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής. Έχουμε τους στόχους του φόρου του 2018, αλλά επίσης αυτή η τοποθέτηση δεν ε, είναι κάτι το οποίο βγαίνει αυτομάτως από το Συμβούλιο Σταθερότητας, από το Σύμφωνο Σταθερότητας μάλλον, και ούτε από την κυκλική οικονομία. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε την ε, ε, Οικονομική Νομισματική Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχουν συμβαστικές λύσεις μεταξύ κρατών μελών και Ευρώπης και έτσι να είναι πιο ανθεκτικές οι οικονομίες μας. Βέβαια, αυτά αφορούν όλες τις δραστηριότητες, την ε, απασχόληση, τις ε, και πρόκειται για προσπάθειες που έχουν απτυχθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά είναι πιο εντατικές πρόσφατα. Κατά την Προεδρία μας θέλουμε αυτά τα θέματα όλα να σημειώσουν πρόοδο. Το δε Σεπτέμβριο έχουμε το ΕΚΟΦΗΝ στο Ταλίν. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε ένα έγγραφο προς συζήτηση και αν εμβαθύνουμε αυτό θα είναι μία μακρόπνη προσπάθεια. Έτσι θα θωρακίσουμε την Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Θα έχουμε και νομοθετικές προτάσεις για επενδύσεις, για τραπεζική ένωση, για την ένωση των κεφαλαίων και άλλα και για φορολογία. Ως Προεδρία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να σημειωθεί πρόοδος για όλους αυτούς τους τομείς, να υπάρξει στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, στενή συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη γνώμη στο εχουμε κάποιε σημαντικέ νομοθετικέ νομοθετικές προτάσεις πρώτα-πρώτα όσον αφορά την επέκταση αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Η νομοθετική αυτή πρόταση είναι πολύ σημαντική και έχει περάσει από διαπραγματεύσεις, επαφές των συνομοθετών. Ξεκινήσαμε από τον τριμερή διάλογο του Μαΐου και είμαι θα ότι οι επαφές, οι συζητήσεις αυτές θα οριμάσουν και θα γίνουν συμφωνία. Αυτό το οποίο θα το προσπαθήσουμε και αύριο που έχουμε τριμερή διάλογο. Οπότε έτσι θα ολοκληρώσουμε ε, αυτή την προσπάθεια όσο γίνεται πιο γρήγορα και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει οι πόροι του δημοσίου τομέα να γίνουν επενδύσεις που είναι αυτό το οποίο χρειάζεται οικονομίας. Επίσης θα πρέπει ε, να δούμε την προτεραιότητα των θεμάτων της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Ε, αυτό επίσης είναι μακρόπνο όραμα. Θα πρέπει να υπάρξει αλληλοκατανόηση των όσων θέλουμε σε διάφορα ζητήματα πολιτικά αλλά και τεχνοκρατικά, τεχνικά. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πετύχουμε και είναι εφικτό να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα πρόοδου και θέλουμε να γίνουν διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, με την ιεραρχία των πιστωτών και έτσι να πάμε σε κάποια θέματα μεταβατικού χαρακτήρα όσον αφορά την ε, επαναξιολόγηση και τροποποίηση ε, της οδηγίας για κυφολογικές απαιτήσεις. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε πάσα δυνατή πρόοδο όσον αφορά την ε, πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Σήμερα στο Συμβούλιο συμφωνήσαμε για ένα κοινό σχέδιο δράση όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Και είπαμε ότι κάθε συμφωνία θα πρέπει να έχει θετικέ επιπτώσει όσον αφορά την κατανομή του κινδύνου και υπάρχουν και συγκεκριμένα μέτρα διαφύλαξης όσον αφορά ε, το, το, τους φορείς εξυγίανσης και όσον αφορά τα μέτρα προστασίας των ε, αποταμιεύσεων. Οπότε και εμείς θα συνεχίσουμε ε, να εργαζόμαστε όσον αφορά την κεφαλαία αγορά. Υπάρχουν μια σειρά προτάσεων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη σταθερότητα αυτών των ε, αγορών και όσον αφορά την Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών. Θέλω συγκεκριμένα να σταθώ τώρα στη βελτίωση της υποδομής. Αυτό ήταν αντικείμενο του σχετικού κανονισμού στις ρυθμίσεις για εποπτεία και στις ρυθμίσεις για εξυγίανση. Επίσης αυτό αφορά και τα συνεξοδοτικά ταμεία. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν, το ώστε το Συμβούλιο να καταλήξει συγκεκριμένε θέσεις το συντομότερο. Η Προεδρία επίση θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξουν κάποια μέτρα σε συνέχεια της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης του προγράμματος δράσης για τις ε, κεφάλαια αγορές. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι οι συνομοθέτες οφείλουν να συμφωνήσουν όσον αφορά την αναθεώρηση της τέταρτης οδηγίας κατά του ξεπλήματος χρημάτων. Αυτό καταπολέμει και την τρομοκρατία είναι επομένως πολύ σοβαρό και για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να έχουμε φιλόδοξα αποτελέσματα και νομικά βιώσιμα. Τέλος, δύο λόγια για μια δίκαιη φορολογία. Αυτό είναι κοινή μας μέρημνα. Τα κέρδη πρέπει να φορολογούνται εκεί όπου γεννώνται, εκεί όπου δημιουργούνται. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η στρέβλωση της αγοράς και να υπάρχει αποτελεσματική ίσπραξη. Μας απασχολεί όλους αυτό. Και όλα αυτά θεωρούνται εκ πρώτης όψεως προφανή. Όμως στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα πρέπει να συγκεράσει κανείς διάφορα ζητήματα δύσκολα από πολιτικής πλευράς και τα κράτη-μέλη γι' αυτό ανησυχούν, για το αν υπάρχουν ίση όροι και συνθήκες. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πρόοδος τεχνολογίας επίσης, αλλά και η διεθνή συγκυρία. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δούμε πώς θα φορολογηθούν οι ολοένα και πιο ε, ψηφιοποιημένες οικονομικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για διάφορα θέματα και έτσι θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό για τον ΦΠΑ τον Νοέμβριο στο Συμβούλιο. Να δούμε τι γίνεται με τις ε, σχετικές δημοσιεύσεις και επίσης τι γίνεται με τη δέσμη μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα εγκρίνουμε ε, κάποια μέτρα για τις μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την πρόταση της Επιτροπής για να θεσπιστεί οδηγία του Συμβουλίου όσον αφορά την ε, φοροαποφυγή και όσον αφορά την φορολόγηση των εταιριών. Επίσης έχουμε την πρόκληση της ε, φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς η γλωσσική και η πολιτιστική πολυμορφία ε, είναι ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μια συνεργασία γεμάτη αλληλοσεβασμό. Να, και το σύμβολο της ε, Προεδρίας μας. Καινοτομία. Κανείς να μην χάσει το τρένο. Είμαστε όσον αφορά την ποιότητα ζωής οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Άρα να εξασφαλίσουμε και σε εμπορική και σε οικονομία ένα ανοιχτό πνεύμα, αλλά και στην κοινωνία μας. Ασφάλεια να κυριαρχήσει σε κάθε τομέα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τόμας, για αυτήν την εξαιρετική παρουσίαση. Συμφωνώ πολύ με τις προτεραιότητες που μας περιέγραψες. Και έχουμε καλά νέα, διότι σήμερα μόλις ψηφίσαμε την πρώτη δέσμη μέτρων Fast Track με την ε, κατεπίγουσα διαδικασία και παρουσιάσαμε τη, τη δεύτερη πρόταση. Θα μπορέσουμε σύντομα λοιπόν να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους μαζί σας σύντομα. Έχω να σας κάνω μια έκκληση. Δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε δύο σημαντικού σε τριμερεί διαλόγους με τη Μαλτέζικη Προεδρία. Ε, το FSI2 και την ε, καταπολέμηση της νομιμοποίηση ε, παράνομων εσόδων. Ελπίζω λοιπόν η δική σας Προεδρία να μπορέσει να δώσει θετική ορμή στα θέματα αυτά Χρειάζεται να βρούμε συμβιβασμού και να ολοκληρώσουμε τα δύο αυτά σημαντικά θέματα. Αυτό είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, διότι χρειαζόμαστε περισσότερε επενδύσει. Είναι σημαντικό όμω και για την ε, καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Δεν θα θέλαμε να κολλήσουν τα θέματα αυτά, θα θέλαμε να προχωρήσουμε. Και βέβαια δεν περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα θέματα αυτά αύριο, είναι όμως σημαντικό να διατηρηθεί η ορμή και να ολοκληρωθούν τα θέματα αυτά. Είναι λοιπόν μια έκκληση προς εσάς. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω την ε, σημασία του τομέα της φορολογίας και επικροτώ αυτό που είπατε. Έχουμε εδώ πέρα ε, τον ε, εισηγητή για την κοινή φορολογική βάση των εταιριών ε, που αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της δίκαιης φορολόγησης αλλά και η στρατηγική για την ενιαία αγορά κεφαλαίων. Πρώτος ομιλητής είναι ο Αντρέας Σβάμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε βρίσκομαι σήμερα εδώ, διότι ο συνάδελφος Μπουρκχαρτ Πάλς δεν μπορεί να είναι παρόν. Ε, χαιρόμαστε που η Εστονία είχε αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον οικονομικό διάλογο στον οποίο αναφερθήκατε κατά την παρουσίασή σας. Αναφερθήκατε στην εμβάνθυνση της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ε, και είπατε ότι ε, θα είναι εδώ θέμα και οι αρμοδιότητες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, η Εστονική Προεδρία τι θα κάνει σχετικά με το θέμα των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών και του ε, Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Και επίσης, πού βρίσκεστε ποια είναι η θέση σας όσον αφορά αυτήν την ευρωπαϊκή ασφάλιση για τους ανέργους και πώς βλέπετε τις συζητήσεις στο Συμβούλιο να προχωράνε. Επίσης, ε, όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της ΕΚΟΝ, ξέρετε ότι το ΕΛΚ υποστηρίζει τη φορολογική διαφάνεια και γι' αυτό είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα πολύ ισχυρή διαπραγματευτική εντολή στο θέμα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιες είναι λοιπόν οι ανησυχίες του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη φορολογική διαφάνεια όπου είναι αυτό απαραίτητο και προσυμφέρον των φορολογούμενων στα κράτη-μέλη. Ε, πρόεδρε, αυτές ήταν οι δύο μου ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση φυσικά είναι πολύ σημαντική και θέλουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της. Σχεδιάζουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό στην άτυπη ε, ε, συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών στο Ταλίν με βάση το έγγραφο του Μαΐου που θα αποτελέσει πολύ καλή βάση. Το ίδιο έγγραφο Ανατολισμού αποτελεί και πολύ καλή περίληψη όλων των προτεραιοτήτων που έχουμε θέσει για τους εαυτούς μας στο εγγύς μέλλον. Καταρχάς, ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και θα πρέπει να ε, ξαναυπάρξει εμπιστοσύνη στο σύστημα και να υπάρξουν ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομικά και οικονομικά στα κράτη-μέλη. Δεύτερον, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα και να ολοκληρώσουμε την ε, Τραπεζική Ένωση. Και όσον αφορά θέματα παρακολούθησης και όσον αφορά ε, και όσον αφορά νομισματικά θέματα και όσον αφορά τον προπολογισμό, ε, είναι σημαντικό να είναι σαφώς καθορισμένες οι αρμοδιότητες των Υπουργών. Και έχουμε καταρχάς τα θεσμικά ερωτήματα. η συζήτηση των θεμάτων αυτών ε, δημιουργεί και νέα ερωτήματα. Και όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο θέλουν οι χώρες της Ευρώπης να προστατεύσουν, ε, να διαφυλάξουν κάθε ευρώ που ξεπερνάει το 1% του ΑΕΠ όταν μιλούν για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. αν αυξηθεί η συνεισφορά τους, ε, τότε ε, ο ρόλος των κρατών μελών θα είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι είναι σήμερα στην Ευρωζώνη. Και όσον αφορά την φορολογία, αναλάβαμε από τη Μάλτα την Προεδρία και θα θέλαμε πολύ να συνεχίσουμε από το σημείο που σταμάτησε η Μάλτα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις εκθέσεις αναχώρα και την ομολογία και την οδηγία για ε, τις κεφαλαιακές απαιτήσει. και η προηγούμενη Προεδρία, η Σλοβακία, έκανε πολλή δουλειά πάνω στο θέμα αυτό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως δεν έχει να κάνει μόνο με την αύξηση της ε, διαφάνειας στην ε, φορολογία. Το συζητάμε φυσικά αυτό, συζητάμε όμως και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αγορά και πώς ερμηνεύουμε τις συνθήκες. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου έχει πολύ σαφή θέση στο θέμα αυτό και πολλά κράτη-μέλη ανησυχούν. Γενικά θα συνεχίσουμε τις εργασίες στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου για να βρούμε λύσεις στις ανησυχίες των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Thank you, Ευχαριστώ, Περβάνς Περές. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, πολύ κουράγιο για την Προεδρία σας. Το δεύτερο εξάμεινο είναι πάντοτε πιο δύσκολο διότι υπάρχει μεγάλη πίεση για να επιτευχθούν αποτελέσματα θα ήθελα να επεκτείνω την ερώτηση του συναδέλφου από το ΕΛΚΑ. Ο καθένας έχει τη δική του θεώρηση, αλλά υπάρχουν θέματα ανησυχίας για μας, ε, τα αναφέρατε ε, στην εισαγωγή σας σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν σας ζητάμε να τα επιλύσετε όλα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, αλλά ε, είπατε για το, το, την άτυπη του Σεπτεμβρίου που θα είναι ένα ραντεβού σημαντικό. Είσαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποια είναι η δική σας θεώρηση για την συνέχεια των σχέσεων μεταξύ Συμβουλίου και, και Κοινοβουλίου. Στον τομέα αυτό είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας. Ε, Βγαίνουμε από μια περίοδο προγραμμάτων σε πάρα πολλές χώρες ε, και είχαμε το πρόγραμμα το δινηρό για την Ελλάδα και είχαμε δομές άτυπες για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε, να παρατηρούμε, να παρακολουθούμε. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα για το οποίο είναι όλο και πιο ευαίσθητοι οι συμπολίτες μας. Στο Συμβούλιο λαμβάνονται αποφάσεις που επιβάλλονται στην εθνική κυριαρχία χωρίς να υπάρχει μια πραγματική συζήτηση, μια λογοδοσία κατά κάποιο τρόπο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι θέμα για το, την Ευρωζώνη αλλά και για το ΕΚΟΦΗΝ, διότι στο ΕΚΟΦΗΝ εγκρίνονται οι συστάσεις αναχώρα. Ε, ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό και έχω μια πιο ειδική ερώτηση ε, για ένα φορολογικό θέμα. Άλλοι συνάδελφοι θα ε, αναφερθούν σε άλλα σκέλη της φορολογίας σχετικά με τον ΦΠΑ, σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είχαμε μια ομοιρία κατά κάποιο τρόπο αυτού του φακέλου που είχε ξεκίνησει καλά με την προηγούμενη Προεδρία. Αλλά ποια είναι τα στοιχεία, ποια είναι η προοπτική κατά τη γνώμη σας, ούτως ώστε να καταλήξει ο φάκελος αυτός, ελπίζω, στην Προεδρία σας, αυτός τον φάκελο τον οποίον περιμένουν αυτοί που ασχολούνται με εκδόσεις, ώστε να υπάρχει ε, θεμητός δίκαιος ανταγωνισμός. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Θα ήθελα να αρχίσω με την τελευταία ερώτηση, τη ηλεκτρονικό βιβλίο και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις. Ασχολούμεθα με το θέμα αυτό και θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο την πρόταση όταν θα είναι έτοιμη ε, και όταν θα έχουν ρυθμιστεί οι διαφορές και θα ήθελα να σας παραπέμψω σε ένα έγγραφο της Επιτροπής που είναι μια καλή βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις αλλά πρόκειται για ένα θέμα πολύ περίπλοκο. Είναι δύσκολο να έχουμε πρόοδο στον τομέα αυτό και να έχουμε σύντομα αποτελέσματα. Ναι, ναι, δεν απαντήσατε στην πρώτη μου ερώτηση. Νόμιζα ότι θα απαντήσετε αργότερα και σχετικά με τον δεύτερο ερώτημα δεν αναφερθήκατε στην ουσία του θέματος. Ο φάκελος αυτός ήταν περίπου έτοιμος και ένα κράτος μέλος ε, το, καπι, καπηλεύθηκε αυτό το φάκελο κατά κάποιο τρόπο. Πώς θα βρεθεί ο πολιτικός ε, δρόμος για να ξεμπλεχθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Αυτό που μπορώ να πω σχετικά με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις είναι ότι το προηγούμενο Συμβούλιο συζήτησε το θέμα, αλλά η ομοφωνία απαιτείται εδώ. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ομοφωνία σήμερα στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Αλλά όπως είπα, εργαζόμαστε για το θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο θα είναι ικανοποιητικό για όλα τα μέρη. Είπα στην αρχική μου παρουσίαση ότι ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας το θέμα αυτό θα κλείσει. Αλλά νομίζω ότι απήντησα στην πρώτη σας ερώτηση. Όχι. Um, Ashley Fox. Ashley Fox. Ε, καλησπέρα κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα ε, να συγχαρώ τη χώρα σας ε, για τις πρόοδους που έχει κάνει στην ψηφιακή ε, καινοτομία και το Gulf Tech είναι νομίζω ένα μοντέλο από το οποίο όλοι μπορούμε πολλά να μάθουμε. Όσον αφορά στις, στα εικονικά νομίσματα, και στην τεχνολογία, η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ και το Γιβραλτάρ είναι μέρος της εκλογικής μου περιφέρειας, άρχισε μια δημόσια διαβούλευση, μια κανονιστική, ένα κανονιστικό πλαίσιο για αυτήν την τεχνολογία. Το πλαίσιο αυτό θα διευκολύνει προοδευτικό περιβάλλον ασφαλές για τις χώρες που χρησιμοποιούν το μέσο αυτό. Και Ελπίζω να συνεργαστούμε με όλες τις εταιρείες που ε, θέλουν ε, να συνεργαστούν στο Γιβραλτάρ. Ελπίζω η χώρα σας να τρέφει συμπάθεια προς το θέμα αυτό. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να μάθει από την προσέγγιση του Γιβραλτάρ η Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν θα προωθήσει η νομοθεσία η Προεδρία σας θα το λάβει υπόψη το θέμα σχετικά με την ε, νομοθεσία περί καινοτομίας. Είμαι εδώ σήμερα ως ε, ε, Προεδρεύων ε, του ΕΚΟΦΗΝ, του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Δεν συζητήσαμε το θέμα αυτό στο επίπεδο του Συμβουλίου. Και νομίζω ότι η ΣΥΝΤΕΚ είναι σημαντικό θέμα και θα έπρεπε να ενταχθεί στον γενικό κανονισμό η Κομισιό υποσχέθηκε ότι στο πλαίσιο της Ένωσης των Κεφαλαιογορών θα υποβάλει πρόταση μέχρι το τέλος του έτους και ελπίζω ότι θα έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε ενδελεχέστερα το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ παρόν στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Είμαι από α, τις κατοχώρες ένας συμπολίτης μου. Αγαπά πάρα πολύ τη χώρα σας και το λαό σας τόσο πολύ ώστε αν, ανέπτυξε μια εκστρατεία εκπληκτική χρησιμοποιώντας όλα... Ε, smartest, uh, rightist, uh, όλα τα... Και γιατί το έκανε αυτό. Το έκανε διότι όλοι σας αγαπάμε στον Ία και επαναλαμβάνω τα όσα λέχθηκαν. Αν είστε ε, από, από χώρα που αρχίζει από ε, οπότε όλα τα electronic θέματα θα τα επιλύσετε και θέλουμε να σας συγχαρούμε για την ψηφιοποίηση περίπου όλων των τομέων και θα ήθελα ε, να θέσω μια ερώτηση για την ΣΥΝΤΕΚ, για την FinTech. Στο Κοινοβούλιο θετήσαμε φιλόδοξη έκθεση και τώρα τελειώνουμε τις ε, διαβουλεύσεις για την FinTech ε, και προετοιμάζουμε το πρόγραμμα δράσης της FinTech το φθινόπωρο ούτως ώστε να διευκολύνουμε ε, την ταχύτατη αντιμετώπιση λόγω των εξελίξεων θα, θα συνηγορούσα όπως και ο συνάδελφος Φόξ να εστιαστούμε ε, περισσότερο σε όλες τις ε, εξελίξεις στην FinTech όχι μόνο για τα εικονικά νομίσματα που είναι σημαντικά για την οδηγία περί ξεπλήματος χρήματος. Θα ήταν καλή ιδέα αν θα μπορούσατε όλο αυτό το πακέτο να το αντιμετωπίσετε την ε, εισήγησή μας και ε, την έκθεση της Κομισιόν στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ αν παρουσιάσει το σχέδιο δράσης Κομισιόν το φθινόπωρο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να έχουμε ένα πλήρες σχέδιο δράσεως με πίνακες για να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα στο επόμενο εξάμεινο suur tänu küsimuse eest ja on väga meeldiv kuulda, et äh, Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να ακούει κανείς ότι υπάρχουν φίλοι, ότι υπάρχει αγάπη για τη χώρα μας και ότι η εκστρατεία ΕΣΤ ήταν τόσο δημοφίλισμα και στη χώρα μου και τα παιδιά μου έλαβαν μέρος σε την εκστρατεία. Πολλοί φίλοι προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε όσο μπορούσαμε περισσότερα για αυτή την καμπάνια ΕΣΤ. Ήταν κάτι που ήταν πολύ πολύ ευχάριστο, κάτι χαρούμενο για τη χώρα. Τώρα, FinTech και ο σχετικός κανονισμός. Ναι, ναι, σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει το θέμα να συζητηθεί στην άτυπη συνοδοκορυφή του Σεπτεμβρίου. Ελπίζω ότι θα έχουμε φρέσκες ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα προωθήσουμε το θέμα. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Δημήτρης Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Εστονία για τα πολύ μεγάλα βήματα στην ψηφιοποίηση και της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης της χώρας σας. Πριν μία εβδομάδα παρουσίασε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τους στόχους της Εστονικής Προεδρίας ο Πρωθυπουργός σας, ο κ. Ράτας. Τον ρώτησα τι σκοπεύει να κάνει η Εστονική Προεδρία για την ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα. Και μου είπε ότι είναι μέσα στις προτεραιότητές σας. Θα ήθελα να μου πείτε πιο συγκεκριμένα πράγματα, πώς σκέφτεστε ο κοινωνικός πυλώνας να αποκτήσει υπόσταση και να μην είναι απλώς μία ετικέτα χωρίς περιεχόμενο. Το δεύτερο θέμα αφορά στα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου στις 31 Μαΐου του 2017 τα υπολογίζει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Τι σκοπεύει να κάνει η Εστονική Προεδρία στα θέματα τραπεζικής εποπτείας πτωχευτικού δικαίου για να μειωθεί το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που στη χώρα μου την Ελλάδα ή στην Ιταλία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Το τρίτο θέμα αφορά στην φορολογική εναρμόνιση που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κραυγαλαίας φοροδιαφυγής. Πολλές πολυεθνικές πληρώνουν πολύ λιγότερους φόρους από ό,τι μισθωτοί συνταξιούχοι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι σκοπεύετε να κάνετε σε αυτό. Και τέλος, άκουσα ότι ε, επιδιώκεται την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης. Εκρεμεί η υλοποίηση του τρίτου πυλώνα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, το EDIS. Υπάρχει μια πρόταση της Κομισιόν, αλλά δεν προχωρά διότι ορισμένα μέλη του Συμβουλίου βάζουν ουσιαστικά εμπόδια σε αυτή την πρόθεση. Χωρίς τον τρίτο πυλώνα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ποιήση. Τι θα κάνει η Εστονική Προεδρία για να προχωρήσει η τραπεζική ενοποίηση και με τον τρίτο πυλώνα. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Καλύψατε σχεδόν όλα τα θέματα στην ερώτησή σας. Αλλά ας αρχίσουμε από το πρώτο νόημα που αφορά τον κοινωνικό πυλώνα. Προς το παρόν ομολογώ ότι δεν έχω ακόμη στοιχεία για το πόσο έχουμε προχωρήσει. Ελπίζω, σας τα είπε πιστικά ο κύριος Ράτα στην Ολομέλεια. Τώρα, όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Από το 2014 το ποσοστό τους συνεχώς μειώνεται. Οι δε, οι Υπουργοί Οικονομικών το εδήλωσαν σήμερα. Εμεί θέλουμε μια πολύπλευρη προσέγγιση. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η εποπτεία. Σημαντικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επ' αυτό. Επίσης, χρειάζεται ένα πρόγραμμα δράσης για να καλύψει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τους επιχειρηματίες. Κατά τρίτον, θα πρέπει να συνεχίσουμε όσον αφορά την πτωχευτική νομοθεσία και να λύσουμε κάποια διαρθρωτικά προβλήματα. Τελευταίο, οι ίδιες τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν τις ε, μεταρρυθμίσεις της λειτουργίας τους. Προτιθέμεθα να τροποποιήσουμε την νομοθεσία ούτως ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος με συγκεκριμένα μέτρα. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Πιστέψτε με, το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά το θέμα και πρόκειται να συνεχίσουμε να συζητούμε στο Συμβούλιο. Πάντως, Ήδη έχουμε τάξει τι προτεραιότητε. Πρώτα όλα είπαμε ότι θα επικεντρωθούμε στο όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων. Οπότε αυτό το νομοθετικό πακέτο είναι προτεραιότητα τη Προεδρία μα. Θέλουμε επίση να συμφωνήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά κάποια επίγοντα μέτρα μείωση ε, των κινδύνων. Και για άλλα μέτρα. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο συμβουλίου. Αυτό είναι το ελάχιστο το οποίο χρειάζεται ούτως ώστε να προχωρήσει η υπόθεση σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Σας τονίζω, θα συνεχίσουμε να ε, προσπαθούμε για την ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης και για το θέμα των καταθέσεων. και πρόκειται να συζητηθούν όλες οι επιλογές που αφορούν αυτό το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Thank uh, Ευχαριστούμε. Περιμένουμε ανυπόμονα τις προτάσεις. Σβέν Γκίγκολτ. Καλώς ορίσατε κύριε. Και οι πράσινοι σας ε, ευχόμαστε. Απλώς επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπαν οι άλλοι συνάδελφοι ότι και εμείς συμμαθούμε πάρα πολύ την ε, χώρα σας και Ξέρετε, έχω αναμνήσεις πολύ ρομαντικές κάποτε που πήγα εκεί διακοπές. Βεβαίως και είναι υπέροχο μέρος να πάει κανείς. Τι, α, είσαι και περίεργος, ε, τι έγινε. Καλά, καλά, θα στα πω μετά, πιούμε μια μπυρίτσα. Πάντως, τώρα στα σοβαρά. Είναι υψηλή προτεραιότητα ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος. Είναι προτεραιότητα μετά από όσα έχουν γίνει και για να τα καταφέρουμε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια σειρά θεμάτων που εκκρεμούν. Δεν τα έχει αντιμετωπίσει το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει κάνει πολλές προσπάθειες όσον αφορά την έρευνα για τα Panama Papers. Θέλουμε να ασχοληθούμε πιο σοβαρά, εις βάθος με το θέμα, ας πούμε όσον αφορά ε, τα υποθηκοφυλακία, τα, τα μητρώα, ε, εσείς είσαστε παράδειγμα προς για την διαφάνεια. Ε, θα ήταν το φυσιολογικό αυτό. Όλες οι χώρες να πασχίζουν για την maximum διαφάνεια. Γιατί είναι ξεκάθαρο τι γίνεται με την κυριότητα της γης και τι γίνεται με τον πραγματικό δικαιούχο άσχετα με την νομική μορφή εκάστης εταιρεία. Ε, άρα αυτό ελπίζουμε να μας βοηθήσει η Προεδρία σας και να έχουμε φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την διαφάνεια τώρα. Και τη φοροδιαφυγή πρέπει να κυνηγήσετε. Να, ακολουθώ το παράδειγμα των φιλελευθέρων, βλέπετε. Και όταν λέμε για καταπολέμηση φοροδιαφυγής, ξέρω ότι έχετε ένα ιδιόμορφο φορολογικό Γιατί ας πούμε για τις εταιρείε έχετε μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Μα πώς θα αποφύγετε αυτό το χρησιμοποιήσουν ε, αλλοδαπή ούτως ώστε να αποφύγουν τη φορολόγηση. Αυτό μας προβληματίζει. Επίσης, Σύντομα, αλλά δύο θέματα. Έχουμε την πρόταση όσον αφορά τους ε, ενδιάμεσους, τους μεσάζοντες και όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα, δυστυχώς, αναβλήθηκε η σχετική απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ. Θα δώσετε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα κατά την προεδρία σας, διότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε επιτέλους. Όπως είπατε, η Εστονία παγίως συμφωνεί με τη Γερμανία όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά. Οπότε έχω και εγώ ένα τελευταίο ερώτημα. Για δώστε μας ένα-δυο παραδείγματα ε, διαφωνία σας, έντονης με τον κύριο Σόιμπλε. Εγώ διαφωνώ μαζί του. Οπότε θα με καθησύχαζε αν και εσείς μου δίνετε παραδείγματα διαφωνία σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κίκολτ. Ενδιαφέρον το ότι θίξατε το θέμα της Γερμανίας. Ε, εγώ έμαθα γερμανικά στο σχολείο μου και πάντα χαίρομαι που μπορώ να μιλώ με τον κύριο Σόιμπλε και τους αυστριακούς συναδέλφους στα γερμανικά. Χαίρομαι επίσης όταν ακούω ε, ανθρώπους να έχουν περάσει καλά στην Εστονία. Υποψιάζομαι κιόλας γιατί το λέτε αυτό. Όσον αφορά τώρα την οδηγία για την ε, καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Αυτό είναι σημαντικό θέμα και για την Εστονική Προεδρία. Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε του τριμερεί διαλόγου όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αύριο θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία να ε, αναλάβουμε συγκεκριμένα βήματα. Η Μάλτα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ε, προεδρίας έκανε πολύ καλή δουλειά στους τρίμερι διαλόγους και με λύπη διαπιστώσαμε ότι το σημαντικό αυτό, η σημαντική αυτή δέσμη μεταρρυθμίσεων, ε, δηλαδή η οδηγία για την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων, έχει γίνει έχει καθυστερήσει επειδή ε, ένα θέμα δεσπόζει στη συζήτηση που είναι η δημοσίευση πληροφοριών. Δεν θέλουμε ασαφείς ή άδικες λύσεις. το Συμβούλιο πιστεύει ότι πρέπει να έχουμε αδιάβροχη νομοθεσία, να το πω έτσι. Ε, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύση, θα πρέπει όμως να εργαστούμε σκληρά. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε συμβαστική λύση, δυστυχώς, ακόμα. Αυτό πάντως είναι σημαντικό στοιχείο της δέσμης μέτρων και σημαντικό είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία στις τροπολογίες. Ο τριμερής διάλογος θα συνεχιστεί αύριο. Και θα ξεκινήσουμε αμέσω τη συζήτηση του θέματος αυτού. Και κατόπιν θα δούμε ποια θα είναι η τελική λύση όσον αφορά τον πραγματικό δικαιούχο και τη δημοσίευση των πληροφοριών. Ε, το Συμβούλιο έχει κάνει ένα μεγάλο ε, βήμα προς την κατεύθυνση του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Όσον αφορά το φορολογικό σύστημα της Εστονίας, ε, θα ήθελα να σας καθησυχάσω. Δεν είναι μηδενικός ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος και είναι 20% όταν παίρνει κανείς χρήματα από την επιχείρηση. Η φορολογική μας βάση είναι ευρεία. Δεν έχουμε τομεακές ή περιφερειακές ρυθμίσεις. Μία η ιδιαιτερότητα είναι ίσως ότι φορολογούμε τα μερίσματα κατά την διανομή τους, κατά την κατανομή τους. Ευχαριστώ. μπορείτε επίσης ε, να μας δώσετε μια σύντομη ερώτηση για τους μεσάζοντες, για τους ενδιάμεσους. Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σχετικά, ε, είναι σχετικά πρόσφατη. Σήμερα μόλις παρουσίασε ε, την πρόταση και θα την εξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Μπάρμαρα Κάπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Χαίρομαι και εγώ που μπορώ να σας μιλήσω γερμανικά. Μας είπατε ότι μιλάτε γερμανικά, ότι καταλαβαίνετε γερμανικά. Ε, την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτώ την Εστονία. Σήμερα δεν μπορώ να σας ε, ε, ε, πω τις εντυπώσεις μου. Τρία θέματα θα ήθελα να αναφέρω από αυτά που, αναφέρατε εσείς. Το ένα είναι η δημοσιονομική πολιτική και η ε, εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα. Τα κράτη-μέλη τις εφαρμόζουν πολύ αργά. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει, θα είναι λογικό να έχουμε κίνητρα για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν καλύτερα τις ε, συστάσεις αναχώρα. Αναφέρατε ότι θέλετε να δημιουργήσετε κίνητρα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και το ερώτημα είναι τι κίνητρα θα δημιουργήσετε ώστε οι χώρες να μπορέσουν να, τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τις συστάσεις ανά χώρα. Δεύτερο θέμα, η φορολογία. Αναφερθήκατε στην ψηφιοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε εδώ και πολύ καιρό εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι επιστώνουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά την ψηφιοποίηση της φορολογίας. Η χώρα σας είναι πολύ προηγμένη τεχνολογικά και ε, θα ήθελα να ρωτήσω τι μέτρα έχετε στον τομέα της φορολογίας και όσον αφορά το ΦΠΑ πώς ε, βλέπετε την πρόταση του Κοινοβουλίου να έχουμε χαμηλότερους συντελεστές ε, για τα ηλεκτρονικά μέσα. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, νομίζω ότι μπορούμε να αναφέρουμε τη καλή πρακτική του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι, όπου ο, αυτός που έχει την πλατφόρμα να είναι αρμόδιος για την ίσπραξη του ΦΠΑ. Τρίτη παρατήρηση, η καταπολέμηση της φοροαποφυγής ε, που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό θέμα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω εδώ μια ερώτηση. Υπάρχουν ε, από τον ΩΣΑ κατευθυντήρες γραμμές, υπάρχει το σχέδιο δράσης για την διάβρωση της φορολογικής βάσης ε, και την μεταφορά κερδών, τον BEPS. Θα πρέπει ε, ως Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα. Η ερώτησή μου προς εσάς είναι ε, πώς ε, βλέπει το ΕΚΟΦΗΝ τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Όσον αφορά την ψηφιακή οικονομία, Θεωρούμε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τον ορισμό της έδρας. Ε, δεν θα πρέπει να είναι η φυσική έδρα ο τόπος φορολόγησης, θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε εικονική έδρα. Και έτσι να ορίσουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις. Η Ευρώπη θα μπορούσε να ηγείται παγκοσμίω στο θέμα αυτό και είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κατά τη διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας καταλήξαμε σε ευρεία συμφωνία πάνω στο κείμενο. Η πρόταση αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στην στρατηγική για την ψηφιακή έννοια αγορά και γι' αυτό είναι στρατηγικά σημαντική και για την Εστονία. Θελήσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία κατά την συνάντηση του ΕΚΟΦΗΝ τον Νοέμβριο. Θα χαρούμε πολύ αν το Κοινοβούλιο μας συναντήσει στα μισά του δρόμου. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στο θέμα αυτό. Οι εισαγωγές, οι επιγραμμικές πλατφόρμες, είναι θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, είμαστε όμως διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις. Έχουμε σχέδια, θέλουμε να υποβάλουμε κάποιες ιδέες. και θα συνεχίσουμε από το σημείο που σταμάτησε η Μάλτα όσον αφορά την κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη εξέταση της πρότασης και θέλουμε να υποβάλουμε κάποιες πρώτες συστάσεις σχετικά με τη φορολόγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ενοποίηση είναι δυνατόν να συζητηθεί μόνο αφού επιτευχθεί η συμφωνία όσον αφορά την κοινή ενιαία φορολογική βάση εταιριών. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι και εγώ που έχουμε αυτήν την ανταλλαγή εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Το Συμβούλιο ενέκρινε μια θέση πρόσφατα για μια γεράρχηση των πιστωτών των χρεωστικών μέσων στα πλαίσια της οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίαση των τραπεζών και μια ταχύρυθμη διαδικασία για, ε, ε, για, το πρότυπο IFRS 9 για την αντιμετώπιση του μεγάλου κινδύνου ε, στα πλαίσια αυτά. Η Προεδρία μπορεί να μας πει πώς σκέφτεται να προχωρήσει σχετικά με τα τμήματα που απομένουν για το τραπεζικό ε, πακέτο, CRD, SRMR. Με συγχωρείτε για τα ακρονίμια. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ως Προεδρία θα θέλαμε να συνεχίσουμε μειώνοντας τον κίνδυνο για τα τραπεζικά ιδρύματα και θέλουμε να εισαγάγουμε νέα μέτρα, μεταρρυθμισμένα μέτρα τα οποία θα εγγυηθούν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους στόχους της. Τα μέτρα αυτά είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης στο επίπεδο των κρατών μελών. Το να βρούμε μια ισορροπία στην εποπτεία και στην, για την ανάκαμψη και εξυγίανση πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο την ε, οικονομία και τις εξελίξεις της και θέλουμε να βρούμε μια αναλογική προσέγγιση. Όταν εφαρμόζουμε διεθνείς συμφωνίες τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ευρωπαϊκές αγορές και τις ιδιαιτερότητές τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω Νομίζω ότι όσα άκουσα από την Εστονική Προεδρία είναι πάρα πολύ καλά, ότι θα αποδώσετε ιδιαίτερη σημασία στην ψηφιακή οικονομία και στο θέμα της φορολογίας. Νομίζω ότι αυτό χρειαζόταν και πρέπει τα θέματα αυτά όχι μόνο να εξεταστούν αλλά και να υπάρξουν δράσεις. Έχω μια διτή ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα για αυτό που θα κάνετε για την φορολόγηση της ψηφιακή οικονομίας παραδείγματο χάρη νομίζω ότι ίσως έχετε ιδέες για το θέμα αυτό κυρίως εφόσον χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι 27 προσεγγίσεις Έχουμε τα διάφορα, τις διαφορές στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, ε, στην Αγγλία. Έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Νομίζετε ότι είναι εφικτή μια κοινή προσέγγιση κυρίως όσον αφορά τα συστήματα εταιρικής φορολόγησης και θα ήθελα Επίσης, να μου πείτε αν εισαγάγεται την φορολόγηση ε, στην ε, ψηφιακή οικονομία. Αυτό είναι καλό πράγμα. Ο Αντελαμασούρ και εγώ, οι συγητές, έχουμε ε, πει ότι πρέπει να υπάρξουν άτομα που να είναι υπεύθυνα ψηφιακά. Οι πλατφόρμες να μην μπορούν να ξεφύγουν. Αλλά θα θέλαμε να δούμε αν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι CC του BB ε, και αν υπάρχει μία κατεύθυνση και όχι δύο κατευθύνσεις. Ευχαριστώ. Αναφέρθηκα ήδη στο θέμα αυτό, απατώντας σε μια άλλη ερώτηση προηγουμένως. Η ψηφιακή οικονομία, η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας έχει ενέχει ζωτική σημασία και όπως είπα προηγουμένως, στο σημερινό κόσμο δεν είναι μόνο ο φυσικός ε, τόπος δραστηριότητας που είναι σημαντικό. Θα πρέπει και να βρούμε εικονικό τόπο δραστηριότητας και να αποφασίσουμε για τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Είναι ζωτικό και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουμε αυτή την οδό όσο το δυνατόν ταχύτερα. Επίσης, ανέφερα το θέμα CCCTB, δηλαδή της κοινή ενοποιημένης εταιρικής φορολογικής βάσης. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η εξυγίανση και η ενοποίηση είναι εφικτή μόνο όταν θα, είναι εφικτή μόνο όταν θα έχουμε επιτύχει μια συμφωνία. Ευχαριστώ. δεν θέλετε να μπείτε σε λεπτομέρειες σχετικά με την πρότασή σας. Επανέρχομαι στο δεύτερο μέρος της ερώτησης που είναι σχετικά απλό. Εισαγάγοντας φορολογία στην ψηφιακή οικονομία μέσα στα πλαίσια της κοινή βάσης ή χωριστά. Ιδαλλιώς θα έχουμε δύο προσεγγίσεις δεν είναι τόσο ένα τεχνικό θέμα όσο ένα πολιτικό θέμα. Σας ευχαριστώ. Ίσως. Θα έπρεπε να σας τα πω σαφέστερα. Ένα πρόβλημα που έχουμε είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν προτίθενται, δεν έχουν οριμάσει όσον αφορά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων φορολογικών. γενικώ και ειδικώ. Η πρόταση όσο έχει σήμερα οδηγεί στο ότι κάποια κρατημέλη έχουν χωρίσει περισσότερες φορολογικές αρμοδιότητες από όσο άλλα κρατημένα. Όμως όλα αυτά προβλέπονται από το CCTV. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας σχετικώς. Γκολτιέρι. σας ευχαριστούμε. Μοργάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Αν κανείς ε, διεξέλθει αυτό το πρόγραμμα της Προεδρίας σας, και σήμερα όπως επιβιώθηκε από όσα μας είπατε προφορικά με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι θέλετε να προχωρήσετε με αποφάσεις για την Τραπεζική Ένωση και για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Επομένως, έτσι θα σταθεροποιηθούν τουλάχιστον καταρχήν ένα χρονοδιάγραμμα και κάποιες αρχές για το επόμενο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τώρα όσον αφορά τα θέματα, όσον αφορά το έγγραφο για την χρηματοδότηση της Ένωσης, λέτε ότι υπάρχει η πρόθεση ούτως ώστε να προχωρήσουμε για να έχουμε τον εξονισμό του ΦΠΑ και λέτε ότι η σχετική προβληματική ε, όσον αφορά του εταιρικού φόρους που μας είπατε στην αρχή ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση όσον αφορά την φορολόγηση της ε, ψηφιακής οικονομίας και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, λέτε, οι διαφορές μεταξύ κρατών ε, μελών. Εγώ επιτρέψτε να σας πω ότι από όσα έχω μελετήσει δεν προβλέπεται πουθενά το να υπάρξει καθολική χρήση των ιδίων πόρων. Αν μπορείτε, πέστε με δύο λόγια παραπάνω. Δηλαδή, πώς εσείς θα υπερκεράσετε αυτές τις διαφορές όσον αφορά τη φορολογική πολιτική. Θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση για τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσον αφορά την ολοκλήρωση της Νομισματικής Ένωσης, εσείς απαντήσατε όσον αφορά ε, τις ε, καταθέσεις και την εγγύηση αλλά προτίθεστε να συζητηθούν οι δυνατότητες του προπολογισμού και για την Ευρωζώνη ο υπουργό. Σας ευχαριστώ για αυτό που ρωτήσατε μάλιστα η Προεδρία μας θα κρατήσει έξι μήνες. Έχουμε εντάξει φιλόδοξους στόχους και θέλουμε να πετύχουμε όσο γίνεται περισσότερο για την Προεδρία βέβαια. Όμως δεν να τα καταφέρουν. Καταλαβαίνετε. Όσον αφορά τώρα τον εξονισμό του ΦΠΑ. Δεν έχω διαβάσει τα κείμενα, δεν μπορώ να σας πω πόσο αξιόλογα είναι τα σχετικά. Ούτε το πιο, ποια θα ήταν η πιο δόκιμη λύση, ούτε το τι είναι πιο σκόπιμο να κάνουμε. Το θέμα βεβαίως και είναι ευρύτερο. Το κατά πόσο χρειάζεται να υπάρξει κοινοτική αρμοδιότητα για τα φορολογικά ή όχι. Από τη μια μεριά κανείς θα έλεγε όχι. Αν ακολουθούσαμε τόσο προβλέπονται, δεν θα χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια και άλλες κοινωτικές πολιτικές που επηρεάζουν την απάντηση που θα έδινε κανείς. Πάντως, γενικώς διαπιστώνουμε ότι πρέπει να γίνει η συζήτηση του θέματος τώρα ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις ε, ας το μελετήσουμε αυτό πολύ σοβαρά Σας ευχαριστώ πολύ Πέστε μας όμως, ε, τι λέτε για τους ιδίους ε, πόρους, πέστε μας τι θα ισχύσει για την Ευρωζώνη. Ε, σύμφωνα με όσα ακούσαμε, έχετε άποψη. Πέστε μας. Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή την ερώτηση. έχει συμφωνηθεί το πλαίσιο για την Ευρωζώνη. Νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να απαντήσει άλλος σε αυτό το ερώτημα και όχι εγώ. Thank you. Uh, on this topic we will need to Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε φυσικά το διάλογο, διότι η Επιτροπή μας έχει οθετήσει διάφορες προτάσεις ε, μεταξύ άλλων για τη δημοσιονομική ικανότητα. Φυσικά είναι ε, δύσκολο το θέμα αυτό και δεν ε, περιμένουμε από την Εστονική Προεδρία να ολοκληρώσει την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση μέσα στο επόμενο εξάμεινο, αλλά ελπίζουμε να κάνετε κάποια βήματα προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζουμε στην επόμενη κοφή να γίνεται αλλαγή απόψεων πάνω στο έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθώ και πάνω σε άλλα θέματα που σχετίζονται με το μέλλον του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι επίσης πολύπλοκο θέμα. Νομίζω πάντως ότι τα δύο αυτά θέματα θα πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Είχατε τη δυνατότητα να αναπτύξετε περαιτέρω τις απαντήσεις πάνω σε κάποια ε, σημαντικά θέματα. Κάποια από αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο όχι προσωπικά, αλλά θα συνομιλήσουν ε, τα δύο θεσμικά μας όργανα αύριο σε τριμερή διάλογο. Ελπίζουμε έτσι να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια βήματα πρόοδου. Και έτσι μέσα στους επόμενους μήνες να σημειώσουμε βήματα πρόοδου και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα που να οδηγήσουν σε περισσότερη απασχόληση και περισσότερη καινοτομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λήξη